η διάταξη προβλέπει πρώτα την εκλογή του Προέδρου. Σύμφωνα με το άρθρο 12, οι αρχαιρεσίες για τον Πρόεδρο και το Προεδρείο προβλέπουν ότι ο προηγούμενος Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του επομένου ή την υποψηφιότητά του η πρώην πρόεδρος ε, είπε ότι είναι διατεθειμένη να ασκήσει την προεδρία με το άρθρα 12 και 16 του κανονισμού και γι' αυτό είμαι εδώ. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίασης. Σας υπενθυμίζω ότι στόχος μας τώρα είναι η συγκρότηση σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου και ενός δύο αντιπροέδρων και κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση εκτός αν αφορά αυτό το θέμα της εκλογές ή την επαλήθευση των διαπιστευουτηρίων. Θα εκλέξουμε λοιπόν πρώτα τον πρόεδρο. Με βάση την προσωρινή προεδρία του προηγούμενου πρόεδρου. Λοιπόν, πρώτα η προετοιμασία. Υπάρχει απαρτία, είναι 13 μέλη απαρτία, διαπιστώνω ότι υπάρχουν του παρόντα 13 μέλη και άρα υπάρχει απαρτία. οι πολιτικές ομάδες ή τουλάχιστον 5% των μονίμων μελών να δηλώσουν υποψηφιότητες, κύριο Σάρκας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βάσει των συμφωνιών που έχουν γίνει μεταξύ των πολιτικών ομάδων και προβλέπει την Προεδρία της Επιτροπής Απασχόλησης από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, η δική μας πολιτική ομάδα θεωρεί ότι η καλύτερη, καλύτερος υποψήφιος είναι η τρέχουσα πρόεδρος, εσείς δηλαδή κυρία Μπερές, και θα ήθελα επομένω να σας προτείνω ως υποψήφια πρόεδρο. Καμία άλλη υποψηφιότης, όχι. Σύμφωνα με το 13.1 δέχομαι την υποψηφιότητα αυτή και έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τα συμφέροντα σύμφωνα με την προσθήκη 1 που υπάρχουν στην ιστοσελίδα επειδή μόνο ένας υποψήφιος υπάρχει, εγώ δηλαδή, πρέπει εννέα τουλάχιστον μέλη να ζητήσουν μυστική ψηφοφορία αν θέλουν, όχι, άρα προτείνω να γίνει εκλογή διαβαής. Εδώ γράφει ότι ο προσωρινός πρόεδρος καλεί τον εκλεγμένο να καθίσει στη θέση του. Ορίστε, το έκανα. Και σας ευχαριστώ για την ανανέωση της εμπιστοσύνης. Τώρα το 3. Εκλογή αντιπροέδρου ή αντιπροέδρων. Και εδώ πρέπει να εκλέξουμε τέσσερις αντιπροέδρους και καλώ έναν έναν τους υποψηφίους για πρώτο, δεύτερο, τρίτο αντιπρόεδρο. Οι υποψηφιότητες από τις ομάδες για να δω ποιοι είναι οι υποψήφοι για πρώτη αντιπρόεδρη. Ποιοι είναι. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Την Νάντια Χέρς να προτείνω σαν πρώτη αντιπρόεδρο από την άλλη. Άλλες υποψηφιότητες δεν υπάρχουν. Η κυρία Νάντια Χίρτς αν θέλει να λάβει θέση της, αυτή τη θέση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και αυτού οι οποίοι κάνουν την πρόταση. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ. Α εκλέξουμε λοιπόν διαβοή στην κυρία Νάντια Χέρς. Και σας καλώ να έρθετε εδώ δίπλα μου, εξεβονίμων. Θα εκλέξουμε δεύτερο αντιπρόεδρο. Υπάρχουν υποψηφιότητες για αυτή τη θέση στην Επιτροπή μας. Προτείνουμε, η ομάδα μου προτείνει την κυρία Ζιμπέρ. Ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Κυρία Ζουμπέρ, συμφωνείτε να αναλάβετε αυτές τις ευθύνες. Έχετε συμπληρώσει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Καλημέρα σε όλους και όλες. Πράγματι είμαι έτοιμη να δεχθώ αυτή την ευθύνη και έχω ήδη καταδιαβιβάσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Σας προτείνω λοιπόν να εκλέξουμε διαβοή στην δεύτερη αντιπρόεδρο Et je vous invite, euh, Madame Zuber, à Κυρία Ζουμπέρ, ελάτε, ελάτε μαζί μας στα προεδρικά εδόλια. Περνάμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου υποψηφιότητες, κυρία Μαρή. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Σωρή. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να προτείνω τον κύριο Τόμας Μάν σαν υποψήφιο που μέχρι τώρα ήταν αντιπρόεδρος να συνεχίσει λοιπόν σε αυτή τη θέση. Άλλη υποψηφιότητα δεν υπάρχει. Τέταρτος υποψήφιος υπάρχει. Κύριε Ορί, ε, θα τα μιλήσετε όχι. Λοιπόν, πού είμαστε. Εκλογή τρίτου αντιπροέδρου της Επιτροπής. Υπάρχει υποψηφιότητα η θέση του τρίτου αντιπροέδρου της Επιτροπής. Η κυρία Λαμπέχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω την κυρία Ελίζα Πεσάτα να πάρει τη θέση τρίτης αντιπροέδρου στην Επιτροπή. Πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο για να υπάρξει ισορροπία των φίλων. Η Ελίζα Πεστρέτερ, λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Λαμπέρ. Κυρία Σρέτερ, συμφωνείτε? Θέλετε να λάβετε αυτά τα καθήκοντα. Έχετε συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Έχω κάνει τα μαθήματά μου, λέει η κυρία Σρέτερ, και είμαι σύμφωνη να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Σας προτείνω διαβόηση να εκλέξετε και την κυρία Σρέντερ. Και την προσκαλώ να έρθει και αυτή στα προεδρικά δόλια. Nous allons donc procéder à l'élection de notre quatrième Τέταρτος αντιπρόεδρος. Υπάρχουν υποψήφοι. Κύριε Ορία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Τόμας Μάνι ήθελα να προτείνω. Επαναλαμβάνω την πρόταση που έκανα και προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Άλλε υποψηφιότητες για αυτή τη θέση. Όχι. Κύριε Τόμας Μάν, συμφωνείτε με την ε, πρόταση αυτή. Έχετε συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Έχω κάνει δημόσια τα οικονομικά μου συμφέροντα και θα ήθελα <laughs> να αποδεχθώ αυτή την πρόταση διότι μέσα στη τριπλική πλειοψηφία των γυναικών ίσως ένας άνδρας μπορεί να βοηθήσει. Προτείνω λοιπόν να εκλέξουμε και τον κύριο Τόμας Μαν με διαβοής. Et je l'invite à rejoindre notre... τον καλό να έρθει εδώ στη θέση μας, στο Προεδρείο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου. Να ευχηθώ καταρχάς πάρα πολύ καλή χρονιά, 2012. Σε πιο ζεστό κλίμα θα μπορούσαμε να το κάνουμε πίνοντας ένα ποτηράκι στο τέλος της ημέρας, εφόσον είναι η πρώτη συνεδρίαση. Είναι πολύ σημαντικό, παρά τις πολιτικές μας διαφορές, για τις οικογένειές μας και για μας και για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά το 2012 που νομίζω ότι θα είναι πολύ πλούσια όσον αφορά τα θέματα που έχει συζητήσει η Επιτροπή μας και θέλω να βασίζομαι σε ένα Προεδρείο τόσο ανισόρροπο από πλευρά ισορροπίας φίλων αλλά εξισορροπημένο πλευρά πνευματικών ικανοτήτων. Να σας πω ότι προφανώς για λόγους ανεξαρτήτως της βουλήσεώς μου οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έχουν ήδη εκδώσει ανακοινωθέν τύπου που ανακοινώνουν τη σύνθεση του Προεδρίου. Δεν καταλαβαίνω πώς τη πρακτική ακολούθησαν, αλλά δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Πάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και προτείνω να το εγκρίνουμε όσε σας διανεμήθη. να σας πω ότι προσθέτουμε ένα σημείο 24α που θα αφορά την ψηφορία για την προφορική ερώτηση για την παρέκκληση για την κρίση του του ΦΕΜ. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, άλλη τροποποίηση. Εγκρίνεται τροποποιημένη η ημερήσια διάθεση. Προτείνω να εγκρίνεται τα πρακτικά της, ε, του Νοεμβρίου. Ο κ. Σωρή θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω κάποια αλλαγή. για το σημείο 26 και το σημείο 27 υπάρχει κάποιο πρόβλημα ερμηνείας θα έλεγα και οι σοσιαλιστές μεταξύ ε, σοσιαλιστών, ΕΛΚ και Προέδρου. Διορίστηκε ε, εμπειρογνώμων από πλευράς του Κοινοβουλίου στο Ινστιτούτο του Τωρίνου. Στα πρακτικά Υπάρχει λάθος στα πρακτικά, λοιπόν. Τον Οκτώβριο ανανεώσαμε αυτόματα τη θητεία αυτού που είχε διοριστεί και εδώ φαίνεται ότι κάποιος υποψήφιος διαφωνεί και δεν θέλει να συνεχίσει. Το Δεκέμβριο επανεξετάσαμε το θέμα, κάναμε μια πρόταση, θελήσαμε να αλλάξουμε τη θέση, το διορισμό αυτού δεν αναφερόταν πλέον η αριστεία, η προσωπικότητα του υποψηφίου. Θέλαμε να αλλάξουμε το σύστημα του τρόπου διορισμού. Θέλαμε πρώην Ευρωβουλευτή να προτιμηθεί τη θέση που είχε εργαστεί σε αυτή την Επιτροπή και γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και γνωρίζει πολύ καλά το Κοινοβούλιο. Άρα είναι σε καλή θέση για τις σχέσεις μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου και του Κοινοβουλίου. Θέσαμε το πρόβλημα ασυμβατότητας το Δεκέμβριο. Δεν διαφάνησαν τέτοια προβλήματα ασυμβατότητας και θελήσαμε να βρούμε πρώην βουλευτή που να καλύψει αυτή τη θέση. Ποιο είναι το πρόβλημα ξανά άνοιξε συζήτηση και δεν ελήφθη απόφαση τον Οκτώβριο για την αυτόματη ανανέωση της θητείας. Δεν ήταν ε, πλήρης η αντιπροσωπεία και βάσει των ιδεών που είχαμε θεωρήσαμε ότι πρέπει να βάλουμε ή πρώην συνάδελφο της πολιτικής ομάδας είτε αν υπάρχει πλειοψηφία που το υποστηρίζει να ψηφίσουμε να συζητήσουμε, ε, ψηφίσουμε αλλαγή του τρόπου διορισμού. Αυτό που αποφάσισαν οι συντονιστές. Ακόμα εκκρεμεί το θέμα, είναι ανοιχτή συζήτηση. Δεν θέλω να δυσκολεύσω τις συζητήσεις, ήδη υπήρξαν προβλήματα κάτω παρελθόν μεταξύ μας. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Πολιτισμένα. Προτείνω λοιπόν να μπει αυτή η ψηφοφορία για αυτό το θέμα στη μέση διάταξη. Ευχαριστώ κύριε Ρή, προτείνεται δηλαδή τροποποίηση της ε, ημερήσιας διάταξης. Ναι, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να προβλέπουμε μία ψηφοφορία για ενδεχόμενη αναθεώρηση των αποφάσεων των συντονιστών. Εν τη αυτή περιπτώση θα πρέπει να εγκρίνουμε νέο σύστημα διορισμού. Συνεπώς, αυτό το άτομο που θα μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Τωρίνου θα πρέπει να είναι πρώην βουλευτής. δεν γνωρίζουν σε αυτή την αίθουσα ότι έχει συμβολική αξία αυτή η θέση. Είναι κάποιο που πρέπει να φροντίζει για τη σχέση μεταξύ του Ινστιτούτου και του Κοινοβουλίου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό το μέλος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Προσπαθήσαμε μέσω άλλων εγγράφων να αλλάξουμε αυτή τη θέση, να δώσουμε δικαίωμα ψήφου σε αυτό το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό δικαιολογεί ότι θα πρέπει να μπει κάποιος ε, βουλευτής σε αυτή τη θέση. Δεν είχα καταλάβει τι, σε τι προτείνατε αλλαγή της σημερινής διάταξη. Για να σας είμαι ευχάριστη, μπορώ να προτείνω, αν συμφωνούν οι συντονιστές και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι των ομάδων, αυτό το θέμα, το διαδικαστικό της διαδικασίας, μπορεί να βρει δύο λύσεις που προτείνω. Πρώτα απ' όλα, είτε το συζητάμε σε συνεδρίαση των συντονιστών, στο τέλο τη ημέρα, είτε θεωρείται σημείο της Ολομέλειας και αυτό το θεωρώ πιο κανονικό, διότι οι συντονιστέ επεξεργάστηκαν πολύ το θέμα και νομίζω ότι τώρα εναπόκειται στους συντονιστέ να βγουν υπόψη τι συζητήσει που έλαβαν ε, στα πλαίσια τη Ολομέλεια επίτροπή και θα πρέπει η Επιτροπή να ξεκαθαρίσει συνθήκε τι οποίε θα προχωρήσουμε στι ακροάσει και ψηφοφορία όσον αφορά του υποψηφίου για το Ίδρυμα του Τωρίνου αύριο. Λοιπόν, σήμερα προσθέτουμε τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα επαληθεύσουμε υπό ποιε συνθήκε θα διορίσουμε τον εκπρόσωπό μα όταν το σημείο αυτό θα, είναι στην ημερήσια, θα μπει στην ημερήσια διάταξη αύριο. Συμφωνείτε? Και όταν φτάσουμε στη συζήτηση του σημείου αυτού. Λοιπόν, να είστε προσεκτικοί, να κινητοποιηθείτε, να είσαστε παρόντες στο τέλος της συνεδριάσεως. Εντάξει, αποφασίστηκε λοιπόν. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης και στις α, ανακοινώσεις. Μεταδίδεται μέσω, στο διαδίκτυο συνεδρίασή μας, όσοι είδηστε. Μετά λάβατε τα πρακτικά των εργασιών της Επιτροπής Απασχόλησης αφορά το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα 3 και 4 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Αυτή η ανακοίνωση είναι στα διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Λάβατε και ανακοίνωση όσον αφορά τι εργασίε τη αντιπροσωπεία μα στην Κοπενχάγη στα πλαίσια τη προετοιμασία τη Δανέζική Προεδρίας 24-25 Νοεμβρίου αυτή η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Να υπενθυμίσω ότι μετά τις εργασίες και ελπίζω τη μια αρμονική συμφωνία στην αυριανή ψηφοφορία θα έχουμε ένα μικρό κοκτέιλ για να γιορτάσουμε τον καινούριο χρόνο και μπορούμε να ευχηθούμε το καλό όρισες στον κύριο Ροκ Πίτερ εθνικό αποσπασμένο υπάλληλο υπεύθυνο για θέματα κοινωνικά και απασχόληση των κάτω χωρών που θα συμβάλλει στην ισορροπία των φίλων της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Καλώς ήρθατε. Ίσως μπορείτε να σηκωθείτε όρθιος για να σας δούμε. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης όπου θα υποδεχθούμε την κυρία Μετ Φρεντέριξεν και την κυρία Κάρεν Χάκετ Ρουπ ε, που εκπροσωπούν την ε, Δανέζικη Προεδρία. Θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο τις εργασίες μας όμως εν αναμονή της αφήξεώς τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, θα ήθελα εξ ονόματος όλων σας να υποδεχθώ την κυρία Κάρεν Άκερουπ, Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης και την κυρία Φρέντριξαν που είναι Υπουργό Απασχόληση στη Δανία. Όπως έχουμε συμφωνήσει, θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Άκερουπ για τις αρχικές της παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει μία ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε μία μισή ώρα στη διάθεσή μας. Αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε για κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο. Και μετά και η κυρία Φρέντεξαν μπορεί να λάβει το λόγο και μπορούμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση ομαδοποιημένη. Φυσικά τα ερωτήματά σας μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπουργό κάθε φορά. Κυρία Κερού, που έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μπορώ να ξεκινήσω αν δεν έχετε αντίρρηση. Κυρία Μπερές, μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να έρθουμε ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα το πρωί. Κάτι στο οποίο προσβλέπαμε ιδιαίτερα. Μας αρέσει πολύ που είμαστε εδώ και μαζί με τη συναδελφό μου, την Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας για την δανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. η στενή συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι φυσικά πολύ σημαντική για μας, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης οι αποφάσεις μας θα πρέπει να σταθμιστούν σωστά σε σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Ως άμεσα εκλεγμένοι από τους λαούς της Ευρώπης, εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχετε μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη στα θέματα αυτά. Η Δανική Προεδρία έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική καμπή για την Ευρώπη και τον κόσμο. Η κρίση μας έχει πλήξει σοβαρά και θα εξακολουθήσει μάλλον να πλήττει την Ευρώπη για πολύ καιρό ακόμα με σημαντικές επιπτώσεις για εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που χάνουν τη θέση απασχόλησή τους και που μπορεί να πιστεύουν και των άλλων πολιτών που πιστεύουν ότι μπορεί να είναι τώρα η σειρά τους. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές που διατρέχουν την ε, εργασιακή μας αγορά και την κοινωνική οικονομία της αγοράς, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές αυτές για μένα είναι καταρχήν ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια κοινωνική ισορροπία. Τα δικαιώματα των εργαζομένων και η εκπαίδευση των εργαζομένων θα πρέπει να προστατευτούν. Είναι αξίες που πρέπει πάντα να προστατεύουμε. <clears throat> Πιστεύω ότι και οι δύο αυτές πτυχές μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στις ε, εξυγχρονισμένες πολιτικές εμπορίου και επιχειρήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσει εργασίας δεν δημιουργούνται μόνο από πολιτικές απασχόλησεις, αλλά και οι πολιτικές είναι πολύ σημαντικές για να υποστηρίξουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε από τις κοινωνικές μας πολιτικές και πολιτικές απασχόλησεις, να εξασφαλίσουμε ότι η εργασιακή μας δύναμη είναι απασχολήσιμη <clears throat> και μπορεί να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες οι οποίες ανακύπτουν. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η κρίση αυτή θέτει πίεση σε αυτούς οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι και οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο μόνιμου αποκλεισμού από την κοινωνία. Η κρίση επίσης έχει πλήξει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Υπάρχουν κίνδυνοι ότι τα όνειρά τους και οι ελπίδες τους για το μέλλον θα διαψευστούν και θα καταστραφούν αν δεν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι οι νέοι θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να δείξουν το δυναμικό τους. Είναι ένα πρόβλημα όμως αυτό και για το σύνολο της εργασιακής, του εργασιακού χώρου. Αν οι νέοι λοιπόν δεν αντιμετωπιστούν με το σωστό τρόπο για να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για το μέλλον, φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμα σημαντικότερες προκλήσεις τα επερχόμενα έτη. Δεν μπορούμε λοιπόν να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά στην Ευρώπη. Κάθε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει τη δική του οδό για να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων. Σίγουρα όμως <clears throat> μπορούμε να ενθαρρύνουμε οι μεν και τους τε και να δώσουμε λύσεις οι οποίες θα είναι επιτυχείς. Από τη δική μου άποψη, σε μια τέτοια εποχή κρίσης, ο σωστός δρόμος είναι να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες και τα προσόντα μας και να επανεκπαιδεύσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται μια τέτοια αλλαγή δεξιοτήτων. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια μεγαλύτερη απασχολησιμότητα των εργαζομένων. Είναι καιρό η Κομισιόν να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων με ένα τρόπο ο οποίος θα δώσει πρωτοβουλίες, μάλλον με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ξέρουμε ότι 75 εκατομμύρια νέων αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται ούτε σε μαθητεία, ούτε σε πορεία εκπαίδευσης, ούτε εργάζονται. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα στην συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα στο ΕΠΣΚΟ το Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ανεργία των νέων μέσα στα εθνικά προγράμματα. Το να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων θα πρέπει να είναι και ένα τμήμα της ε, άτυπης συνάντησης των Υπουργών ε, απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων και επίσης ένα αντικείμενο της συνδιάσκεψης για την νεολαία τον Απρίλιο. <clears throat> και θα ήθελα, το ελπίζω, να δω εκπροσώπους και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν την συνδιάσκεψη στη Δανία τον Απρίλιο. Στην τρέχουσα χρονική στιγμή θέλω να αναφέρω επίσης ότι το έτος 2012, όπως ξέρετε, έχει καθοριστεί ως το έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργό γύρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων. Μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό το να δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στο να κρατούμε τους ηλικιωμένους στη δουλειά όταν έχουμε τόσους νέους άνεργους. Αλλά ελπίζω ότι ακούγοντας αυτά τα οποία έχω να σας πω σήμερα, δεν θα έχετε καμία αμφιβολία ότι η Δανική Προεδρία και εγώ προσωπικά θέτουμε μεγάλη έμφαση στο να μπορέσουν οι νέοι να περάσουν σε εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση για να είναι στην αγορά εργασίας. Αυτό όμως δεν είναι μια κατάσταση αντιθετική. Πρέπει ενώ παροτρύνουμε τους ηλικιωμένους να εργάζονται, να δώσουμε και κίνητρα και δυνατότητες για τους νέους να είναι στην αγορά εργασίας. Σε ένα όχι τόσο απομεμακρυσμένο μέλλον θα χρειαζόμαστε όλους που θα μπορούν να εργαστούν στην αγορά εργασίας γιατί αυτό μας δείχνουν οι δημογραφικές τάσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητής στη συνεργασία με το Συμβούλιο και εσάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην ακούσετε από μας πάντα αυτά τα οποία θέλετε να ακούτε, αλλά θα σας μεταφέρουμε τη θέση του Συμβουλίου και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις απόψεις σας και να τις μεταφέρουμε στους συναδέλφους μας μέσα στο Συμβούλιο. Θέλουμε να είμαστε μια ανοιχτή και διάφανη Προεδρία και με εσάς και με τους άλλους συνομιλητές μας. Γι' αυτό <clears throat> θα ήθελα να σας αναφέρω ποια είναι τα ντοσιέ τα οποία θα μας απασχολήσουν στο επόμενο εξάμεινο. Ένα σημαντικό θέμα για μας είναι το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η Κομισιόν θα προτείνει μια οδηγία για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας περί αποσπάσεως εργαζομένων και την ε, αντιμετώπιση καταστάσεων οι οποίες έχουν διαμεθοριακό χαρακτήρα. <clears throat> Εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις πρέπουσες και ορθές συνθήκες εργασίας και για τους εργαζομένους αλλά και προς όφελος των εταιριών. Η απόσπαση των εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο έτυχε πολλή συζήτηση και πολλών διαφωνιών και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουν οδηγήσει σε συναισθηματικές αντιδράσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων των κρατών ε, μελών και μέσα και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για τις προτάσεις που θα προέλθουν για τα θέματα αυτά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλε οι προσδοκίε. Να είμαι ακόμα πιο ειλικρινή για να σα πω ότι εάν επιμείνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να εκπληρωθούν όλε οι προσδοκίε του, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Εξ ονόματο τη Προεδρία, εμεί τονίζω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αν το επιτύχουμε όμω, θα πρέπει να βρούμε κοινό έδαφο. και αν μπορούμε να έχουμε συμφωνία επί των αρχών, η λεπτομεριακή εργασία θα είναι πιο εύκολη. Να σας αναφέρω τι πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτό το κοινό έδαφος. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι το θετικό, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και είναι επίσης και ένα σημαντικό ατομικό δικαίωμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά δεν έχει μεγάλη αξία η ελεύθερη κυκλοφορία αν δεν συνδέεται με σωστέ συνδίκε τη εργασίας και αξιοπρεπή αμοιβή. Πρέπει λοιπόν να συμβαδίζουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμεί. Θα πρέπει να καλωσορίσουμε τους εργαζόμενους και τι εταιρείε από άλλα κράτη-μέλη με ανοιχτές αγκάλες. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά όλους αυτούς του εργαζόμενου. Αν όμω οι ξένες εταιρείε αποσπούν συμβόλαια σε βάρος των εχωρίων εταιριών και εργαζομένων, δεν μπορεί κανείς να αναρωτιέται γιατί κάποιες ομάδες του πληθυσμού και κάποιες πολιτικές παρατάξεις αποκτούν μια σκεπτικιστική στάση και εχθρική στάση ενάντια της εσωτερικής αγοράς. Πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει να στραφούμε εναντίον των μη εντύμων εταιριών, των εταιριών μαϊμούδων ή εταιριών γραμματοκιβωτίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για πραγματικές εταιρείε το να εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή για την απόσπαση εργαζομένων. Πιστεύω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Το να μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτό το κοινό έδαφο σε συγκεκριμένε δράσει μπορεί να μην είναι εύκολο, το γνωρίζω. Αν θέλουμε όμω να προχωρήσουμε, ιδίω σε μια εποχή κρίση όπω ανέφερα, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το επιτύχουμε. Πρέπει να δείξουμε στου λαού τη Ευρώπη ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας είναι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικών Θεμάτων. Βάσει της στρατηγικής Ευρώπη 2020 πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο μιας Ευρώπης η οποία θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον οικονομικό και εργασιακό τομέα, ιδίως ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας απασχόλησης. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για αυτό το θέμα μέσα στην κυβέρνηση της Δανίας, επομένως οι διαπραγματεύσεις θα είναι στα χέρια άλλων συναδέλφων. Ως Προεδρία όμως η Δανία θα προσπαθήσει να επιτύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο για τα θέματα αυτά. Τα σχέδια είναι να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα είναι ρεαλιστικό να συμπληρωθούν οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Δανικής Προεδρίας. Τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικά συμπληρώματα στις εθνικές πολιτικές. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν με ένα σωστά στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η προσέγγιση αυτή ισχύει επίσης και για τι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην προκοσμιοποίηση. <clears throat> Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις το Φεβρουάριο με στόχο να επιτύχουμε στο δυνατόν περισσότερη πρόοδο. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι υπάρχει η πρόταση για την ε, για την ε, μεταρρύθμιση των κανόνων του EMF. Εμείς θα εργαστούμε μαζί σας και μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η κατάλληλη προστασία των εργαζομένων. Ένα καλό πλαίσιο εργασίας είναι ε, απαραίτητη βάση για την εργασιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και ένα σημαντικό στοιχείο για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική αλλαγή και τη γύρανση της εργασιακής δύναμης. Η Πολωνική Προεδρία στο Συμβούλιο, μέσα στο Συμβούλιο έχουν προωθήσει πάρα πολύ το έργο για την εκπόνηση μιας νέας οδηγίας. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε μια κοινή προσέγγιση στο Συμβούλιο που θα έλαβε χώρα στο ΕΜΣΚΟ. Εγώ γνωρίζω τώρα η Κομισιόν είναι έτοιμη <clears throat> να προχωρήσει και να κάνει περαιτέρω προτάσεις για να περατωθούν οι διαπραγματεύσεις. Με τον τρόπο αυτό θα επιληθεί το θέμα αυτό. Περισσότερος χρόνος όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθυστερήσουμε και θα βραδιπορήσουμε σε σχέση με τις προσπάθειες αυτές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Είναι σημαντικό για μένα λοιπόν να εξασφαλίσω ότι θα υπάρξει μια ισορροπημένη λύση το θέμα αυτό σας έχει απασχολήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ένα πράγματι πολύ ένα εξόχως τεχνικό θέμα. παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξη για τις δυνατότητες επιτυχίες ακόμα και αν έχουμε αρκετό δρόμο να διατρέξουμε. Ελπίζω ότι από κοινού θα επιτύχουμε στις προσπάθειές μας και προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία μαζί σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα στην Δανική Προεδρία να κλείσουμε το θέμα αυτό. Αυτές ήταν επομένως όχι ακριβώς λίγες, αλλά εν πάση περιπτώσει εναρκτήριες παρατηρήσεις μου. Όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, πριν από λίγες μέρες όταν ξεκίνησε η Ιδανική Προεδρία, είπε ότι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα πάνω από τα ταραγμένα νερά για τους επόμενους έξι μήνες. Ελπίζω ότι όλοι από κοινού θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη εισήγηση που ήταν πολύ αισιόδοξη για την Προεδρία σας. Θα δούμε στο τέλος τι αξιολόγηση θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα σας θέσουν ερωτήματα οι συνάδελφοι. Πρώτα όμως θέλω να δώσω την ευκαιρία και στην κυρία Κάρνα Γαλούπ να παρουσιάσει το πρόγραμμα ή το όραμα της δανικής προεδρίας. Αγαπητοί κύρια Περές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είχα την ευχαρίστηση να γνωρίσω μερικά σας μέλη στη συνάντησή σας στην Κοπενχάγη, στο Υπουργείο και το βράδυ φάγαμε όλοι μαζί πολύ καλά. Και τώρα ανταποδίδω την επίσκεψη ερχόμενη εδώ. Προσβλέπω στη συνεργασία μας τους επόμενους μήνες. Καλή ήταν η αρχή. Είχαμε μερικές πρώτες θετικές συνεννοήσεις προς όφελος όλων των Ευρωπαίων ελπίζω. Όπως είχα πει και τον Νοέμβριο γνωρίζω καλά το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας ιδιαίτερα. Με την τρέχουσα κρίση οι ευθύνες μας πολλαπλασιάζονται. Η επίτευξη των στόχων μας τους επόμενους μήνες δεν θα είναι κάτι εύκολο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα εργαστούμε όσο σκληρότερα γίνεται, αλλά υπολογίζουμε και στη δική σας βοήθεια και υποστήριξη. Όπως είπε και η συναδελφός μου, η Υπουργός Απασχόλησης, η Δανία αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια κρίσιμη περίοδο. Η οικονομική κρίση έχει πολλές, πολύ αρνητικές επιπτώσεις για πολλούς Ευρωπαίους. Άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους ή φοβούνται ότι θα τις χάσουν. Είναι πράγματι πρόκληση αυτό και πρόβλημα. Πολλοί έχουν φτάσει στην απόγνωση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για όσους θεωρούν ότι δεν έχουν πια κανένα μέλλον. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε όλο και περισσότερους να φεύγουν από την αγορά εργασίας. Γιατί καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και αυτό είναι πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάσταση αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την απασχόληση και θα κάνουμε κάτι γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η Πολωνική, Δανική και Κυπριακή Τρόικα θεωρεί τις δημογραφικές απρές προκλήσεις ως κοινή προτεραιότητα. Στον κοινωνικό ιδιαίτερα τομέα θα προσπαθήσουμε πρώτον να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη γιατί τους χρειαζόμαστε όλους. Δεύτερον στην αγορά εργασίας και τρίτον ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες. Πρέπει βέβαια να κάνουμε μερικές επιλογές και να κρατηθούμε γερά από τις κοινέ αξίες της Ένωσης. Το δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες οι νέοι στην Ευρώπη έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση. Εκατομμύρια νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι άνεργοι και ανειδίκευτοι. 35% έχει φτάσει η ανεργία και υπάρχει ο κίνδυνος ολόκληρη γενιά να χαθεί λόγω αυτού. Αυτό πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, διότι γνωρίζουμε και από προηγούμενες κρίσεις ότι όσο πιο πολύ διαρκεί η κρίση, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει κανείς μια δουλειά. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προετοιμάσουμε το μέλλον. Όπως λέει και η έκθεση του κυρίου Θωμά Μαν, οι άνω των 60 θα αυξηθούν τρομερά οι αριθμοί τους. Ιδιαίτερα το 15 με 35 θα αυξάνεται η ηλικιακή αυτή κατηγορία κατά 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ευκαιρία των υπερηλίκων αυτών να παραμείνουν ενεργοί. Θέλουμε να συνεχίσουν να, συμφέρουν, να συμβάλλουν ενεργά στη ζωή της κοινωνίας. Η Δανική Προεδρία θα υποβάλει τα πρώτα της συμπεράσματα για αυτό το δημογραφικό πρόβλημα. Λαμβάνοντας υπόψη και το ότι το 2012 είναι το ευρωπαϊκό έτος για την ενεργή τρίτη ηλικία. Τρία νομοθετήματα κυρίως θα φροντίσουμε. Πρώτον, το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία. Δεύτερον, η οδηγία κατά της άνησης μεταχείρισης και τρίτον, οι αλλαγές στον κανονισμό για το συντονισμό της κοινωνικής πολιτικής possible Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινωνικές αλλαγές και την καινοτομία. Περιμένουμε την έκθεση της κυρίας Στάνοχλ κατά τα τέλη Μαΐου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την οδηγία ίσης μεταχείρισης, συνεχίζοντας τις προσπάθειες της Πολωνικής Προεδρίας και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο για τις αλλαγές προς το καθεστώς, τα κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε μία πρώτη έκθεση του κ. Τσάπανεκ που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ψηφιστεί τέλη Φεβρουαρίου στην Επιτροπή σας. Μαθαίνω. Επίσης θα, συνεχίσετε, θα συζητήσετε και σήμερα το πρώτο σχέδιο αυτής της έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να σας κάνω μία σύνοψη των συναντήσεων που προβλέπουμε και ορισμένων σημαντικών ημερομηνιών. Δύο επίσημες συναντήσεις της ΕΠΣΚΟΡ θα οργανωθούν και μία άτυπη στη Δανία τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα Ιωθώτα, θα αναφέρουμε όλες μας τις προτεραιότητες σε συνεντεύξεις. Το 12, όπως γνωρίζετε, θεωρείται Ευρωπαϊκό Έτος ενεργών υπερηλίκων. Η Δανική Προεδρία θα κάνει μία πρώτη, έκανε ήδη μία πρώτη διάσκεψη περί αυτού την περασμένη εβδομάδα και θα οργανωθεί διάσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού. Στις 5 και 6 Μαρτίου διάσκεψη για, τους, ε, για την απασχολησιμότητα των αναπήρων. Καλέσαμε τον κύριο Κάσα στην διάσκεψη και χαίρομαι που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Στη διάσκεψη αυτή ο κύριος Κόσα θα μας παρουσιάσει την έκθεση ιδίας πρωτοβολίας του για την απασχολησιμότητα των ε, αναπήρων και είναι και πρόεδρος της ε, σχετικής διακομματικής ομάδας στο Κοινοβούλιο. Περιμένω την παρουσίαση και την έκθεσή του. Η Κομισιόν επίσης θα παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση της για την αναπηρία κατά τα τέλη του 12. Επίσης θα αντιμετωπίσουμε και την άτυπη συνάντηση των Υπουργών ΕΠΣΚΟ στις 19 και 20 Μαρτίου στην Κοπενχάγη θα μιλήσουμε για το θέμα της ανέχειας των παιδών και μία προσέγγιση οικογενειακή του προβλήματος. Στις 22 Μαρτίου η ετήσια διάσκεψη για τους Τσιγκάνους, η Ρώμα. Η Δανική Προεδρία και η Κομισιόν θα οργανώσουν τον Απρίλιο μία διάσκεψη μετά την επίσημη συνάντηση των Υπουργών ΕΠΣΚΟ για την απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνικά προβλήματα και ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας. Η ενδέκατη συνάντηση των ανέαπτωχών και ανέργων στις 11 Μαΐου με συμμετοχή ε, ανθρώπων που έχουν ζήσει την ανέχεια με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους. Όσοι ζουν στην ανέχεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ειδικά. Η συνάντηση αυτή οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Ανέχειας. Όπως η συνάδελφός μου υπουργό Απασχόλησης, νομίζω και εγώ ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κρίση και είναι άρα πολύ πιο σημαντικό από ό,τι ποτέ να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και Αναμένω με ανυπομονησία προσδοκώ την ανάληψη δράσης. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Σας είχα υποσχεθεί ερωτήσεις. Θα έχετε 14. Δεν ξέρω αν θα οδηγήσει σε τόσο ζωηρή συζήτηση όπως αυτή που διεξήχθη μαζί σας το δείπνο, το οποίο θυμόμαστε με μεγάλη ευχαρίστηση αλλά θα έχουμε ομάδες τεσσάρων ερωτήσεων, μετά σας δίνουμε το λόγο για να απαντάτε. Ξεκινούν τα δύσκολα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα ξεκινήσω το χρονόμετρο για να ελέγχω πόση ώρα θα μιλάτε. Η πρώτη που θα δώσω το παράδειγμα είναι η κυρία Ράπτη και μετά η κυρία Ραμπέρ. Καλημέρα. Ευχαριστώ τις δύο υπουργούς που είναι εδώ μαζί μας. Τις συγχαίρω διότι μας περιέγραψαν πάρα πολύ ωραία την κατάσταση που υπάρχει. Ε, πέραν όμως από την πολύ καλή περιγραφή, αυτό που θα ήθελα είναι να μας περιγράψουν το ίδιο ωραία και με ακρίβεια τις πρωτοβουλίες που σκοπεύουν να πάρουν πρώτον για να ενισχυθεί η απασχόληση και να καταπολεμηθεί η ανεργία και δεύτερον για την καλύτερη λειτουργία και την αποδοτικότερη λειτουργία του Κοινωνικού Ταμείου. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι εκτός από τους νέους που είναι μέχρι 25 ετών και εκτός από τους μεγαλύτερους που είναι από 60 χρονών και πάνω, υπάρχουν οι εργαζόμενοι που είναι από 25 μέχρι 60 χρονών. Εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της κρίσης. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις, έχουν δάνεια. Νομίζω ότι θα πρέπει και για αυτούς να υπάρχει μέρημνα. Θα ήθελα να ακούσω τις πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε. Γιατί μας μιλήσατε για το τι θα κάνει το Κοινοβούλιο, αυτό το ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά, είμαστε στο πλευρό σας, αλλά χρειαζόμαστε και εσάς να έχετε ισχυρή φωνή στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λαμπέρ και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε επί των στόχων που έχετε θέσει. Αλλά όσον αφορά τι τοποθετήσει, δεν αναφερθήκατε στους εποχιακού εργαζόμενους και τους, ε, τις μεταφορές προσωπικού μεταξύ επιχειρήσεων που είναι πολύ σημαντικό ίσω εργάζονται στον κοινωνικό τομέα, τον τομέα της απασχόλησης. Δικαιώματα στη θέση εργασίας, ε, κοινωνικές ασφαλίσεις είναι σημαντικές πτυχές αυτού του ζητήματος. Πώ συμμετείχατε, με ποιο τρόπο στη συζήτηση μα αυτά τα θέματα. Δεύτερον, αυτή η Επιτροπή σήμερα και αύριο θα συζητά την έκθεση για την επισκόψη της ετήσιας ανάπτυξη, ετήσια επισκόψη για την ανάπτυξη. Σε ανταπόκριση της εκθέσεως που συνέταξε το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημα ρόλο σε αυτόν τον τομέα, αλλά είναι σημαντικό, πιστεύουμε, για τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και για δημοκρατική συμμετοχή να παίξει ρόλο το Κοινοβούλιο. Θα μας ενδιέφερε λοιπόν να δούμε πώς θα λάβετε εσείς υπόψη της ε, τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κάτι που μας απασχολεί, ότι αυτή η έκθεση ανάπτυξης απομακρύνεται τους στόχου του 2020. Επηρεάζεται πολύ από τον οικονομικό προγραμματισμό, επηρεάζεται λιγότερο από τον κοινωνικό προγραμματισμό η Ιδανική Προεδρία τι θα κάνει για να επαναφέρει την ισορροπία όσον αφορά τι απόψει του Συμβούλου για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ η κυρία Χάρκιν και μετά η κυρία Γιασλοβεύσκα. Κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την παρουσίασή τους, πολύ ενδιαφέρουσα. Η παρουσίαση έχω κάποιες ερωτήσει. Έχουμε το Ταμείο Παγκόσμιου. Όπω είπατε προλίγου, η Ευρώπη είναι σε ταραγμένα ύδατα, πλέει σε ταραγμένα ύδατα. Και αν το δει κανείς σε αυτή την πλευρά, θα μπορούσε να αναρωτηθεί τι προτάσεις έχει η Προεδρία όσον αφορά α, την παρέκκληση που προβλέπεται την κρίση. Το Κοινοβούλιο σχεδόν ομόφωνα υποστήριξε το να συνεχιστεί η εφαρμογή ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την εξαίρεση, για την κρίση και ξέρουμε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που ε, μπλοκάρει τις εργασίες. Το Δεκέμβριο 13 χώρες ε, έκαναν αίτηση να ενταχθούν σε αυτή την παρέκκληση για την κρίση. Άρα χρειάζεται αυτό το μέτρο και είχαμε και τρεις, τρία μέλη της Ολλανδίας που ήταν από εκείνους που μπλόκαραν την πρόταση. Εσείς τι προτάσεις έχετε για να προχωρήσει το όλο θέμα. Και η νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνει και τους αυταπασχολούμενους και τους ε, αγρότες. Ποια είναι η υποψή σας. Μετά αναφερθήκατε στην κοινωνική αλλαγή και στην καινοτομία και προτίθεται να κάνετε κάποιες ε, ε, προσπάθειες, κάποιες εργασίες αφορά το πρόγραμμα για, progress, για τη μικροχρηματοδότηση. Τι άποψη έχετε. Μόνο εννέα χώρες έχουν πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και στο σχετικό πρόγραμμα. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό το μέτρο. Πώς μπορεί να συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Είπατε ότι θέλετε να ξαναμπούν οι νέοι στην ε, εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Πολύ καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να βρουν δουλειά στο τέλο του κύκλου. Υπάρχει σχετισμό των δύο πτυχών που ανέφερα. Τέλος αναφερθήκατε στον τομέα τη πρόνοια και της φροντίδας ε, και πώ η μοντέρνα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα. Έχετε κάποιε πιο συγκεκριμένε ιδέε μας σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Γιαζοβιέσκα Και η κυρία Τουρίνεν που εκπροσωπεί τη Δανία. Θα ακολουθήσει η κυρία Γιαζοβλεύσκα. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω προς τις δύο υπουργούς. Πρώτα απ' όλα απευθύνομαι προς την Υπουργό Απασχόλησης. Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Δανέζικης Προεδρίας, δύο ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μας. Η Ευρώπη που είναι υπεύθυνη και η Ευρώπη που είναι δυναμική. Μια Ευρώπη που είναι υπεύθυνη είναι αυτή που θέλει να παγιοποιήσει τα οικονομικά, να ε, στηρίξει, ε, μειώσει το έλλειμμα. Δυναμική Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία επενδύει ε, στα προσόντα των εργαζομένων και αυξάνει τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Το μεγαλύτερο δυναμικό της Ευρώπης είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο οι νέοι. Ποιο είναι το πρόγραμμα της Προεδρίας για να μπορέσει να συνδέσει τους μακροπρόθεσμους στόχους Τη χρηματοδοτικής πολιτικής με του αρχιπρόθεσμου στόχους για την απασχόληση. Τι μπορείτε να κάνετε για να εφαρμόσετε καλύτερα τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει προβλέπεται για το ταμείο αυτό 25% από τα ιδιωτικά ταμεία για την ώρα. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ποια θα είναι η συμμετοχή του κοινωνικού ταμείου στα ιδιωτικά ταμεία Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει. Πρόκειται για μεγάλα ποσά. Αλλά ακούστηκαν κάποιες επικρίσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Πώς μπορεί να αυξηθεί αυτή η αποτελεσματικότητα της χρήσης των κοινωνικών ταμείων, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την κατάρτιση, ούτως ώστε η κατάρτιση να οδηγεί στην απασχόληση. Μετά η κοινωνική ένταξη. Ένα από τα προβλήματα των μέτρων λιτότητας ε, είναι ότι υπάρχει μείωση των δαπανών για την κοινωνική πολιτική. Χρειάζεται να αλλάξουν ε, οι προτεραιότητες. Μεταξύ των προτεραιοτήτων σας, κυρίες μου, βρίσκεται και το θέμα των δίκαιων ε, συνθήκων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ισοτήμων συνθήκων. Κατά την άποψή σα, ποια είναι η πολιτική για κοινωνικές επενδύσεις για να πετύχετε τους στόχους που αναφέρατε. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να πω μια λέξη ακόμα. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο θα επεξεργαστείτε. Κάποια έγγραφα. Διακόπτη η Πρόεδρος. Η κυρία Τούρινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι αν, μπορώ να, αν πρέπει να μιλήσω αγγλικά ή δανέζικα, θα μιλήσω αγγλικά για να με καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι χωρίς διερμηνία. Για την ανεργία των νέων. <coughs> πρέπει να κατανοήσουμε, πιστεύω, ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν είναι στο ύψος του προβλήματος, της διάστασης του προβλήματος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν δείτε την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν για την Ανεργία των Νέων, αν δείτε την ε, ε, διαπίστωση του προβλήματος και μετά τα προτινόμενα μέτρα είναι σαν να πετάει κανείς βότσαλα στη θάλασσα και να περιμένει ότι έτσι θα τη μετακινήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς κάποια πιο στεναρά συμπεράσματα σε επίπεδο Συμβουλίου που θα προωθήσουν το θέμα αυτό λίγο περισσότερο, να υπάρξει ένα σύστημα εγγύησης για τους νέους, κάποιος στόχος απασχόλησης μέχρι το 2020 να υπάρχει κάτι περισσότερο από τα μέτρα που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής. Δεύτερον, για την απόσπαση των εργαζομένων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ένα θέμα το οποίο έχει και συμβολικό χαρακτήρα και πάρα πολύ πολιτικές αποχρώσεις. Θέλω να σας θέσω το εξή ερώτημα. Φαίνεται <clears throat> ότι η Κομισιόν, ότι η θέλει να εξασφαλίσει και κάποια αστική ευθύνη σε επίπεδο πέραν των εθνικών συνόρων. Έχετε κάποια σχόλια σε σχέση με αυτό. Και επίση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στι 9 Δεκεμβρίου είχαν κάποια ανησυχητικά στοιχεία γιατί οι εταιρείε με λιγότερο από 250 εργαζομένου θα έπρεπε, σύμφωνα με την ε, απόφαση του Συμβουλίου, να έχουν ένα πιο ελαφρύ καθεστώ σε σχέση και με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο. Θα σας δώσω το λόγο και στις δύο είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο κάθε <clears throat> ερωτών κανονικά έπρεπε να θέσει μονάχα ένα ερώτημα, αλλά βασίζομαι στην ικανότητά σας να είσαστε συνθετικές και να απαντήσετε σε περισσότερο από ένα άτομο κάθε φορά. Σας δίνω, λοιπόν και στις δύο το χρόνο. Και μετά έχουμε δύο γύρους ακόμα ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στην μητρική μου γλώσσα, επειδή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα αυτά και ελπίζω ότι θα μου δώσει λίγο περισσότερο χρόνο η Πρόεδρος για να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι πολλαπλά τα ερωτήματα τα οποία πηγαίνουν σε πολλές κατευθύνσεις. η ελάφρυνση του διοικητικού άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό σε μια εποχή κρίσης να συζητήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας, να απογραφικοκρατικοποιήσουμε τις διαδικασίες μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των συνδικών εργασίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή που να έχουν απευθυνθεί στο Συμβούλιο και προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το διοικητικό άχθος, αλλά όπως είπα πριν, όχι σε βάρος των συνδικών εργασίας και των συνδικών διαβίωσης των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα σημείο αρχής για μας. Και θα δείτε στα έγγραφά μας ότι το τονίζουμε αυτό σαφώς. Ως χώρα που ασκεί την Προεδρία, δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω έγγραφα τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή ακόμα ένα επίσημο χαρακτήρα και τα οποία είναι αποτελέσματα οικοτολογιών. Επομένως, <clears throat> εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας κανένα τέτοιο επίσημο κείμενο. Επίσης χαίρομαι για το γεγονός ότι μιλάμε για την ανάγκη μεγαλύτερης υπευθυνότητα και πιο μεγάλου δυναμισμού στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα συνθήματα της Δανικής Προεδρίας. Αυτό είναι και το αποτύπωμα που θα ήθελα να αφήσει στην ε, ιστορία της Ευρώπης η Ιδανική Προεδρία. Είναι απαραίτητο να εδραιώσουμε τη μακροοικονομική μας προσέγγιση αυτόν τον γεγονός. Είναι εξίσου σημαντικό όμως το να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα είναι βιώσιμο το ευρώ. Εφόσον πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματά μας, αυτό είναι σημαντικό, αλλά πρέπει παράλληλα να ενισχύσουμε και την απασχόληση και να εξασφαλίσουμε και ότι και η απασχόληση στην Ευρώπη θα είναι βιώσιμη. Τώρα, για το μέλλον είναι κάτι που πρέπει να επιληφθούν του θέματος αυτού όλες οι προεδρίες. Έχετε δίκιο γι' αυτό. Όταν συνεδριάσει το Συμβουλίο την επόμενη Δευτέρα, πιστεύω ότι θα είναι κυρίως το θέμα της απασχόλησης και της ανάπτυξης που θα είναι τα κύρια θέματα συζήτησης. Εγώ πιστεύω ότι εδώ και πολλούς μήνες συζητούμε τα θέματα σε καθαρά μακροοικονομικό επίπεδο. Αλλά έχει σιγά σιγά αναδυθεί μια κοινή συνείδηση ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της περιστολής των ελλημάτων και της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία των νέων, να είμαστε λοιπόν όσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε, ενώ συγχρόνως θα αντιμετωπίσουμε και τα άλλα στρώματα του πληθυσμού, τις άλλες ηλικίε. Δεν υπάρχουν μονάχα οι νέοι άνεργοι, υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι άνεργοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι σε σύνταξη. Σε ό,τι αφορά την αργία των νέων, ότι εμείς θα πρέπει να δώσουμε κάποιες εγγυήσεις στους νέους. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί σε κάθε χώρα σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για να λύσει το πρόβλημα της ε, ανεργίας των νέων. Για μας θα πρέπει ο καθενέας να έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε μια καλή κατάρτιση για τέσσερις μήνες το, το ελάχιστο <clears throat> για το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν μπορώ από μόνη μου να προκαθορίσω το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μειοψηφία εμπλοκή στο Συμβούλιο που εμποδίζει να λειτουργήσει καλά αυτός ο μηχανισμός, που εμποδίζει <clears throat> να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως αυτό το μηχανισμό. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να εργασόμαστε πολλές φορές σε άτυπο επίπεδο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύσεις. Και αυτό ενδεχομένως θα συνεχίσει και στο μέλλον. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο όμω στο μέλλον είναι να σκεφτούμε περισσότερο για το θέμα του κατά πόσον και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Και επίσης θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα των εποχιακά εργαζομένων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης για αυτούς οι οποίοι στις πολυεθνικές εταιρείε μετακομίζουν από μία θηγατρική σε μια άλλη θηγατρική υπάρχει μια ευρεία συνένεση μεταξύ μας ότι θα πρέπει να υπάρχει, αν όχι μια εναρμόνιση, τουλάχιστον μια προσέγγιση της συνθεσίας των εποχιακά εργαζομένων και σε ό,τι αφορά την υποδοχή ειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε αυτούς τους εργαζόμενους. Να μην υπάρχει dumping σε σχέση με τις αποδοχές τους. Όσοι έρχονται από άλλες χώρες θα πρέπει να καλύπτονται ακριβώς από τις ίδιες συνθήκες όσο αυτοί που εργάζονται στις χώρες μας ήδη. Ξέρω ότι κάποιοι θα το επικρίνουν αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο για την εποχιακή εργασία. Για τους ε, νέους αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Δίνει τις δυνατότητες και φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε για την εξισορρόπηση της ε, ζήτησης και της προσφοράς στον τομέα της εργασίας. Τέλεια. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, κύριε Χάγκερ. Ευχαριστώ για όλα σας τα ερωτήματα, εξαιρετικά όλα. Και τονίζουν ακριβώς το θέμα που πρέπει να λύσουμε. Γιατί η Ευρώπη υποφέρει και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γιατρευτεί και να έχουν δουλειά όλοι και όλες για τη στρατηγική του 20 Εμείς αναλαμβάνουμε την Προεδρία τη στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει τόσο μεγάλα προβλήματα. Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην στρατηγική του 2020. Η τωρινή κατάσταση περιγράφεται στην ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την Ανάπτυξη. Δεν είναι πολύ ευχάριστο ανάγνωσμα. Εκεί βλέπετε ποια είναι τα μακροοικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα της απασχόλησης. Και οι τρεις παράγοντες που αναφέρονται εκεί είναι σημαντικοί και πρέπει να τους πάρουμε υπόψη μαζί. Να μην ξεχνάμε ότι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα είναι κάτι σημαντικό. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Η κοινωνική πολιτική δεν είναι απλώς η βοήθεια που χορηγούμε στον κόσμο για να βρει μια δουλειά γιατί ξέρουμε και από την περασμένη δεκαετία ότι έχει τύχει πολλών επιθέσεων. Το Φεβρουάριο το Συμβούλιο θα συζητήσει τα μηνύματα που θα μας δώσει η κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας του 2020. Για την μικροχρηματοδότηση αυτό θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις μετά τη διάσκεψη για τη κοινωνική καινοτομία. Μόνο επί ένα χρόνο υπάρχει αυτή η μικροχρηματοδότηση και πρέπει να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση και να δούμε τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι θετικό, αλλά τα συμπεράσματα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Επίσης έγινε ένα ερώτημα για τις κοινωνικές αλλαγές και την καινοτομία. Και το νέο αυτό πρόγραμμα, η νέα προσέγγιση, θέλει να προσθεθεί ευελιξία με βάση πραγματικά στοιχεία. Το πρόγραμμα θα εξεταστεί στην ομάδα εργασίας για τα κοινωνικά προβλήματα την Άνοιξη. Όπως ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα αυτό σχετίζονται με το πολιετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ξεπερνάει την Προεδρία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Θα σας πω ποιοι ζήτησαν το λόγο για να προετοιμαστούν. Madame Blinkevichute, Madame Sinclair, mm, Monsieur Thomas Mann, puis Monsieur Christensen. Monsieur... Ο κύριος Στέφανος Χιούγκς πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την κυρία Φρέντριξεν ρωτώ. Είπατε στην εισήγησή σας για την ανεργία των νέων ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αλληλοβοηθηθούν τα κράτη-μέλη. Αλλά θα είδατε από τα ερωτήματα ότι πολλούς μας ανησυχεί ο μακροοικονομικός ζουρλομανδίας που επιβάλλεται στα κράτη-μέλη ιδιαίτερα την εξάμετρο. Γιατί ακούγονται ήδη στοιχεία από την Κομισιόν που δείχνουν ότι μόνο η λιτότητα εφαρμόζεται. Ευτυχώς η Δανική Προεδρία λέει ναι μεν λιτότητα αλλά και πράσινη ανάπτυξη και αύξηση της απασχολησιμότητας. Θέλω να μας πείτε πώς θα το κάνετε αυτό στην πράξη και αν νομίζετε ότι υπάρχει κανένα πρότυπο που να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. με πολύ κυρία Μπλίνκαβιτσουτέ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ τις δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις τους. Μέσα στην εργασία σας <clears throat> για, τα επόμενα, για τους επόμενους έξι μήνες έχετε να αντιμετωπίσετε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη και που επηρεάζει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τα μέτρα λιτότητος τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη και τα οποία πλήττουν κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν τις χαμηλότερες αποδοχές. Θεωρείτε ίσως ότι η διαδικασία της μεθόδου ανοιχτή συνεργασίας θα ήταν η πιο πρόσφορη για να εξασφαλίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει και μια συνεργασία για την αντιμετώπιση της ε, ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ο πιο απλός τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την ε, φτώχεια είναι το να έχει μια θέση εργασίας, μια πηγή εισοδήματο. Αλλά αυτή είναι μια ιδανική, ιδεατή περίπτωση γιατί δεν μπορεί ο καθένα πάντα θα έχει μια θέση απασχόλησης. Μήπως όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με το να υπάρχει μια οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως πρέπει να μας αντιμετωπίσει αυτό και ένα θέμα για την Υπουργό Απασχόλησης. Εγώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας σε σχέση με την απασχόληση των νέων και επίσης την απασχόληση των ηλικιωμένων. Αλλά πιστεύω ότι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την απασχόληση θα πρέπει να είναι η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Ξέρω ότι αυτό έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα σαν καθημερινή πραγματικότητα στην Δανία. Είσαστε έτοιμοι να μας διαβεβαιώσετε ότι θα επιστήσετε και την προσοχή των εταίρων σας για το θέμα αυτό. Η κυρία Σενκλέρ και μετά ο κύριος Τόμας Η κυρία Σενκλέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Α, πρώτα κυρία Σανκλέρ, κύριε Μάν. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμά σας ε, επανειλημμένα έχει αναφερθεί. Ε, μάλλον από το Βερολίνο, το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιστήκα. Ο πρόεδρο ο πρόεδρος Επιτροπή Μπαρόσο είπε στο Στασβούργο ότι κάθε μικροσία επιχείρηση είναι μια θέση Εάν δημιουργούσε μια θέση, θα εξαλειφόταν η ανεργία στην Ευρώπη. Καταλαβαίνει η Προεδρία ότι οι υπερβολικέ ρυθμίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφει τελικά καταστρέφουν στι εργασία. Η Ομοσπονδία των Μικρομεξών Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούσαν, παρακαλούν να μην υπάρχει άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρησιμοποιούνται από κοινωνικέ πολιτικέ και μόρφε απασχόληση. Η καταστροφή των επιχειρήσεων και η δημιουργία των επιχειρήσεων καταστρέφονται από αυτέ τι πολιτικέ. Κάποιε περικοπέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μείωσαν τι δημόσιε υπηρεσίε, μείωσαν του μισθού και έφεραν το χάο στη ζωή των ανθρώπων. Συμφωνώ. Πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητε κατάρτιση των νέων. Αλλά είναι απλώ ρητορικό σχήμα αυτό, χωρί συγκεκριμένε προτάσει. Και συμφωνώ με την ενεργογύρανση. Πώ τετραγωνίζεται ο κύκλο όμω. Από πού θα προέρθουν οι θέσει απασχόληση, θα δημιουργήσετε θέσει εργασία δημιουργώντα χιλιάδε ε, προγράμματα κατάρτιση, ε, πίνοντα το αίμα των, των φορολογουμένων. Και, και τώρα είναι το αφέλη του ευρώ σαν νόμισμα. Απέριψαν δύο φορέ, ε, ο λαό απέριψε δύο φορέ το ευρώ. Δεν πιστεύει το ευρώ ο πληθυσμό σα, όπω και ο δικό μα τέλος της δεκαετίας του 90 έγινε εκστρατεία φόβου. Μας είπαν ότι θα χάσουμε θέσεις εργασίας αν δεν είμαστε στο ευρώ. Μείναμε εκτός στο ευρώ και εταιρείε όπως η Nissan παρέμειναν. Απλώς ήταν φοβέρες αυτές. Δημιουργούνται εκτός της ευρωζώνης οι θέσεις απασχόλησης και όχι εντός της ευρωζώνης. Ο κ. Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που έχω. <clears throat> Έχω την εντύπωση ότι η Ιδανική Προεδρία με τις ε, δυναμικές υπουργούς της έχει μια πάρα πολύ δυναμική και σημαντική ε, δυνατότητα να επηρεάσει τα πράγματα στον τομέα τον εργασιακό και το, τα θέματα της ε, απασχόλησης γιατί υπάρχει το μοντέλο της ευέλικτης ασφάλειας το οποίο όπως η κυρία Κρίστενσεν έχει λειτουργήσει πολύ καλά στη Δανία τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την ισότητα των γενεών και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Λοιπόν, το θέμα τη εγγύηση για του νέου, να μπορούν να έχουν ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχουν μια κατάρτιση, αν δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασία, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω ήδη πληροφορήσει ένα Έχω πάρει ερωτήματα από νέου για το θέμα αυτό. Τι μπορείτε να του απαντήσετε, τι δικαιώματα έχουν σε αυτά τα θέματα, με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να του δώσετε κίνητρα. Όχι μόνο οι επιχειρήσει θα πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει και οι κρατικοί φορεί να δίνουν τέτοιε ευκαιρίε στου νέου. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε πραγματικά μια ευκαιρία στου νέου και όχι να λέμε κάπου θα πρέπει να υπάρξει μια ευκαιρία κτλ. Πώ θα το κάνουμε αυτό στην πράξη. Ο καθένα ξέρει ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει το να γίνουν πραγματικά εγγύησεις από το δημόσιο τομέα. Μπορούμε όμως να ζητήσουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο, να υπάρχουν οι ε, ευκαιρίες για τους νέους. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ένα σημαντικό τρόπο να δείξουμε ότι η Ευρώπη πράγματι θέλει να δώσει τις ευκαιρίες προς τους νέους γιατί οι νέοι είναι πράγματι πάρα, έχουν πολύ πιο ενθουσιασμό και κίνητρα από ό,τι από τους γονεί τους κυρία Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την, τις ε, δύο υπουργούς για την παρουσία τους και να τους ευχηθώ κάθε καλή τύχη κατά τη διάρκεια της Ιδανικής Προεδρίας. Πιστεύω ότι τα πράγματα ξεκινάνε καλά για το μέλλον. Να επανέλθουμε στο θέμα, στο μοντέλο της ευέλικης ασφάλειας, όπως ανέφερε ο κύριος Τόμας Μάν. Στο έντυπο EU Observer ελέγχθη ότι αυτό μπορεί να είναι και η λύση για τα προβλήματα που έχουμε, δηλαδή μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασιακή δύναμη. Πολλές χώρες θα ενδιαφερόντουσαν για το μοντέλο αυτό της ε, Δανίας, της ευέλικης ασφάλειας. Αν ίσχυε και στις χώρες αυτές αυτό το μοντέλο, μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπήρξαν μιμητές της Δανίας. Δεν υπήρξε θέληση και από άλλες χώρες να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Θεωρείτε εσείς ότι μπορούμε να πείσουμε σύντομα κάποιες χώρες μέλη να αποδεχθούν και να επενδύσουν στο μοντέλο αυτό, να υπάρχει ένα σύστημα υποστήριξης των ανέργων, ώστε ακόμα και αν δεν έχει κανείς μια θέση απασχόλησης, να έχει ελάχιστες αποδοχές οι οποίες θα μπορούν να βοηθούν και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων αυτό που είναι άνεργοι για να επανέλθουν στην ενεργή αγορά εργασίας. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, εάν υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο όχι μόνο την ευελιξία προωθεί αλλά και την ασφάλεια, τότε θα μπορούμε να έχουμε εξασφάλιση της ευελιξίας. Όσον αφορά το δίλημα που θέσατε, για του ηλικιωμένου που θέλουν παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό και ταυτόχρονα να έχουμε και του νέου που δεν έχουν δεξιότητε, είναι άνεργοι και ακόμα και αν έχουν δεξιότητε δεν μπορούν να βρουν θέση. Διότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργία. Είναι ένα δίλημα, αλλά ένα δίλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η κρίση που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη ε, δεν θα πρέπει να γίνει μάχη μεταξύ των γενναιών, να μην μετατραπεί σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το έτος της ενεργού τρίτης ηλικία και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών εστιάζεται στην αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να λύσουμε την κρίση στην Ευρώπη με μια γενιά, με ένα τμήμα του πληθυσμού που θα πολεμάει το άλλο. Θα πρέπει να σεβαστούμε το ότι οι ηλικιωμένοι έχουν οικοδομήσει τι κοινωνίε στι οποίε ζούμε, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι οι νέοι θα μπορέσουν να έχουν μια εκπαίδευση και μια δουλειά όταν τελικά ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να πολεμά ένα τον άλλον. Θα πρέπει ο... να αναλάβουμε ευθύνε για τον άλλον και να αντιμετωπίσουμε σαν σύνολο την κρίση. Και γι' αυτό αποκαλείται το έτος αυτό έτος αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και ενεργού γύρανσης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει διαμάχη, πρέπει να λύσουμε όλοι μαζί για όλους μας την κρίση. Τόσο αφορά το θέμα της ενεργού γύρανσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπογραμμίσω ότι κάποια από τα καλά πράγματα για την ενεργό τρίτη ηλικία είναι ότι μπορούν επιμακρότερο να προσέχουν να φροντίζουν τους εαυτούς τους οι άνθρωποι αυτοί. Όχι μόνο μπορούν να μείνουν στην αγορά εργασία οι πιο ηλικιωμένοι, αλλά να ζουν και καλύτερα, να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο, καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Και αν τους δίνουμε κατάρτιση αντί μόνο περίθαλψη αν τη χρειάζονται, μπορεί να δώσουμε περισσότερη ελευθερία του το τρόπος να διευθύνουν τη ζωή τους, να μην εξαρτώνται από βοήθεια. Αλλά η βοήθεια που θα παράσχουμε μπορεί να είναι απάντηση στο ερώτημα της κυρίας από την Αγγλία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, άμα σκεφτούμε την τεχνολογία για την πρόνοια και να είναι καλή αφετηρία να το προωθήσουμε αυτό, την τεχνολογία στα πλαίσια της ενεργού της και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ε, απασχόληση επίσης εντός των συνόρων μας. Πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες όλους. Και τώρα στην Ευρώπη δεν δίνουμε ευκαιρίες στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Πρέπει να το εξεργαστούμε αυτό. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όπως αναφέρθηκε. Είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον κόσμο για να ζουν καλύτερα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που, για το οποίο θα μεριμνήσει η Προεδρία. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Θα είμαι σύντομη αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας να έχουμε υπόψη μας την αρχή ότι αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Η καταπολέμηση της ανεργίας αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε κάθε χώρα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία για ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Και μαζί μπορούμε να καθορίσουμε στόχους. Παραδείγματος χάρη, στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 υπάρχει ένας στόχος για μια ανεργία κάτω από το 6%, 5,7%. Και θέλουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Και πέραν αυτού πρέπει να δούμε και ποιες είναι, ποια είναι η εμπειρία της Δανίας όσον αφορά αυτό το θέμα. παρατίθεται και αναφέρεται πολύ συχνά το δανέζικο μοντέλο, αλλά υπάρχει ανεργία μεγάλη και στη Δανία. Και εμείς έχουμε υποφέρει από την κρίση. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Και θα πρέπει να προσέξουμε τα προβλήματα την περίοδο της κρίσης, αλλά μην τα θεωρούμε όλα ότι είναι πάντα μόνο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε θετικά την οικονομία και τις δαπάνες. Είναι σημαντικό αυτό. να βασιστούμε στην πράσινη οικονομία, την καταπολέμηση της ένδυας. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτούς τους τομείς. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε βήματα προόδου. Μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στην πράσινη οικονομία, Φερρυπίν. Όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, προφανώς, θα πρέπει να αποταμιεύουμε περισσότερα χρήματα, ούτως ώστε και σε εποχή κρίσεως να μπορεί να εφαρμόζεται η σωστή πολιτική, ο σωστός προϋπολογισμός. Είμαστε πολύ φιλόδοξα Προεδρία για την πολιτική του κλίματος και εκεί μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα. Υπάρχουν δυνατότητες, μπορεί να συμβεί σε αυτό το τομέα. Μετά στο ερώτημα της κυρίας Σενκλέρ για το ευρώ. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα σωστά το ερώτημα, όμως σαν χώρα που είναι στην Προεδρία και που ανήκει στη, στο ευρώ, είναι κοινή ευθύνη αυτή να κάνουμε να δουλέψει το ευρώ, να μπορεί να λειτουργήσει το ευρώ. Είναι τεράστια ευθύνη αυτή. Είναι προϋπόθεση αυτή να επιβιώσει το ευρώ για να βγει από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά μιλάμε για την ασφάλεια. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Στη Δανία ήταν πολύ σημαντικός παράγων αυτός σέβομαι το γεγονός ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη ποικίλει. Όμως, βλέποντας όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν την ανεργία που ετέθησαν, πρέπει να πω ότι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι να τους εγγυηθούμε καλή κατάρτιση. Επαρκή κατάρτιση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους, να τους εκπαιδεύσουμε. Αυτό είναι ο τρόπος για να βγούμε από την κρίση. Αυτό είναι σημαντικό και για τους νέους και για εκείνους που είναι εκτός αγοράς εργασίας επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τελευταία ομάδα ερωτήσεων και δίνω το λόγο καταρχάς στον κύριο Γκουτιέρες μετά την Αντιπρόεδρο κυρία Νάντια Ο κύριος Γκουτιέρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και έχετε εστιάσει ένα μεγάλο μέρος των παρεμβάσεών σας στα θέματα της ανεργίας των νέων και ελπίζω το εξάμεινό σας αυτό θα είναι πολύ παραγωγικό και καρποφόρο στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η πολιτική δημιουργίας απασχόλησης παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών και αν δούμε μονάχα απομονωμένα αυτήν την ε, πολιτική, υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση, για τη μαθητεία των νέων κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί η πρώτη πολιτική η οποία οδηγεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι η οικονομική πολιτική και η πολιτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε δει ότι πέφτουμε όλο και περισσότερο σε μία ύφεση πηγαίνουμε προς μια χαμένη δεκαετία σε οικονομικό επίπεδο που θα είναι και μια χαμένη δεκαετία για πάρα πολλούς νέους. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, να μην υπάρξει μια απώλεια δεκαετία για τους νέους, χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για αυτά που γίνονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά της εργασίας. Αυξάνεται ο χρόνος απασχόλησης χωρίς να αυξάνονται οι αποδοχές, μειώνονται τα κοινωνικά δικαιώματα, χάνεται το δικαίωμα σε συλλογικές συμβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν τι αντίκρισμα έχουν. Δεν μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα μας βγάλει στην, ε, από την κρίση όταν υπάρχουν πολύ διαφορετικά δικαιώματα των εργαζομένων και πολύ διαφορετικές υποχρεώσεις. Επομένως εγώ συμφωνώ με το να υπάρξει μια εγγύηση προς τους νέους. Αυτό το οποίο δεν αποδέχομαι είναι να υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια επισφαλή σχέση εργασία. Πρέπει το καθεστώς αυτό για τους νέους να είναι χρήσιμο, δηλαδή να δίνει μια σωστή παιδεία και μια σωστή ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και πρέπει να είναι και αξιοπρεπές αυτό το σύστημα, το οποίο σημαίνει πραγματικές αξιοπρεπείς αποδοχές και κοινωνικές εισφορές και παροχές. Πρέπει να έχει και ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα γιατί αυτή τη στιγμή που τα κράτη-μέλη έχουν πολύ λίγα κονδύλια να επενδύσουν, θα πρέπει να λειτουργήσει και η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα αυτό. Κυρία Χίρς και κυρία Ζούμπεα μετά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χίρς. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τον τόπο, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσετε τα θέματα αυτά που καταδεικνύει και τη δέσμευσή σας για την επίτευξη μιας λύσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε στην ανεργία των νέων και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην στρατηγική της Ευρώπης 2020. Θέλουμε να μειώσουμε και το ποσοστό της σχολικής αποτυχίας και αποχώρησης από την εκπαίδευση. Φυσικά είναι αυτό το θέμα το οποίο είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά είναι και ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει και κάποια έμφαση και κάποια πίεση ώστε να ε, μπορέσουν ώστε να, να υπάρξει μια παρότρεση προς τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Επίσης υπάρχει το θέμα της κινητικότητας. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία αγορά και να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη εξίσωση συνθήκων, θα πρέπει να ευνοήσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά είναι πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια προσκόμματα όπως είναι η χρήση των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπάρχουν πάρα πολλές οι αιτήσει των ε, εργαζομένων, των πολιτών μας που θέλουν να εξασφαλίσουν την ευκαιρία να εργαστούν σε μια ξένη χώρα που βρισκόνται και πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, με τη μεταφορά των συντάξεων, με την αντιμετώπιση της ανεργίας κτλ. Τίθεται λοιπόν και εδώ το ερώτημα, μπορείτε εσείς να σκεφτείτε τρόπους να τονώσετε περισσότερο την κινητικότητα των εργαζομένων, να φτιάξετε ένα σύστημα όπου υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία είναι πράγματι διακινούμενα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούν να προσαρμόζονται κάθε φορά σε ένα διαφορετικό από τα 28 συστήματα. Πώς θα υποστηρίξετε την κινητικότητα λοιπόν. Η κυρία Σουμπέρ, η νέα αντιπρόεδρος μας, κάνει την παρθενική τη λοιπόν παρέμβαση. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία μέσα στην Επιτροπή μας. Και μετά ο κύριος Θέρκα θα έχει το λόγο. Κυρία Ζούμπερ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει και με την πορτογαλική πραγματικότητα. Τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια συνάρμοση της πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με την πολιτική λιτότητα και αυστηρότητα που πιστεύω ότι είναι υπερβολική ε, από τα κοινοτικά όργανα και ιδιαίτερα σε χώρες σαν την Πορτογαλία όπου υπήρξε παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την Ευρωπαϊκών Οργάνων. Ξέρουμε ότι η Πορτογαλία βρίσκεται σε μια πορεία ύφεση και θα είναι σε πορεία ύφεση το 2012 κατά 3,7%. Με τις συμφορίες που έχουν γίνει με τα ευρωπαϊκά όργανα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα υπάρξει διευκόλυνση των, απολύσεων στους εργαζο... για τους εργαζομένους θα αυξηθεί η... ο χρόνος εργασίας χωρίς να υπάρχει περισσότερη αμοιβή, θα μειωθούν οι αποσημειώσεις απολύσεως κτλ. και θα υπόκεινται σε πιο δυσμενείς συνθήκες οι εργαζόμενοι. Το ερώτημα είναι, εφόσον εμείς λέμε ότι θέλουμε να ευνοήσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γιατί διευκολύνουμε τις απολύσεις. Γιατί θέλουμε να θέσουμε τα άτομα να εργάζονται σε δυσμενέστερες συνθήκες και να εργάζονται ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν ευνοεί τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικές λιτότητος και η δημιουργία θέσεων απασχόληση δεν μπορούν να συνάδουν. Θα ήθελα όμω να έχω την άποψη των υπουργών, των κυρίων υπουργών για τα θέματα αυτά. Ο κύριο Σέρκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία, στις δύο κυρίες Υπουργούς για τις παρουσιάσεις του σήμερα και για την υποδοχή που μας επεφύλαξαν στην Κοπενχάγη. Έχετε προκαλέσει πολλές προσδοκίες όπως ξέρετε και έχουμε πολλές ελπίδες από τη Δανική Προεδρία να οδηγήσει σε μια πραγματική αλλαγή στο τομέα της κοινωνικής Ευρώπης. Αναφέραν οι συναδελφοί μου σοσιαλιστές ποιες είναι οι Θα αναφέρω και να αναφερθώ και στα σεμινάρια που προβλεπόταν να γίνουν στην Κοπεχάγη 28-29 Ιουνίου που έχει κάπως, μάλλον φαίνεται ότι θα βγει από την ατζέντα, γιατί η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτά δεν είναι καμία επένδυση, αλλά είναι μονάχα δαπάνες και δεν αξίζει να γίνουν τέτοια σεμινάρια. Βρισκόμαστε σε μια τεράστια βιομηχανική κρίση, κρίση απασχόλησης. Η Κομισιόν έχει βγάλει μια πράσινη βίβλο για την αναδιάρθρωση και την μετακίνηση των επιχειρήσεων μετά από δέκα πράσινες βίβλους και πάρα πολλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, τώρα μία νέα πράσινη βίβλος η οποία τα ανατρέπει όλα αυτά. Αλλά κυρίως πρέπει να θυμηθείτε τι έγινε και στην, στο τι είπε και η η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι η ύφεση θα ακυρώσει όλες τις προσπάθειες λιτότητας. Όλα αυτά τα οποία γίνουμε δεν θα οδηγήσουν σε τίποτα, θα είναι μια τρύπα στο νερό, εάν δεν υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό σκέψης, που είναι ουσιαστικά σαν να λέει ο γιατρός κάντε αφέμαξη στον άρρωστο που έχει φθήσει η ε, ευλογιά ή κάτι τέτοιο, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Όχι, δεν μπορεί να λυθεί έτσι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία διακυβεύονται είναι τεράστια. Υπάρχει τεράστια πρόβλημα ανεργίας, αύξησης της, ε, Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που γυρίζουμε 50 χρόνια πίσω. Όλα αυτά σημαίνουν λιγότερες κοινωνικές παροχές, λιγότερη ε, απασχόληση και αυτή τη στιγμή, όταν μόνο σε οικονομικό επίπεδο αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Ευρώπης, δεν πρόκειται να βρούμε κάποια λύση. Ο κύριο Όρη και μετά ο κύριο Κάσλερ, αλλά μετά κλείνουμε και θέλω και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Κύριε Όρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε τις κυρίες Υπουργούς και εγώ. Θα ήθελα να πω ότι και η εισαγωγή και οι απαντήσεις στις πρώτες ερωτήσεις μου δημιούργησαν κάποια κατανόηση και τρέφω κάποια συμπάθεια προς αυτά που άκουσα. Δεν μπορεί μια Προεδρία να λύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά μπορεί να επικεντρωθεί επί προτεραιοτήτων. Ακούσαμε τις προτεραιότητες. Να κάνω μια παρατήρηση. Μιλήσαμε πολύ για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στο ότι είναι θέμα των κρατών μελών αυτό. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αντιμετώπιση ανεργίας, αλλά αλλάζει πολύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε τα διάφορα μέτρα όπως το six-pack ε, που ανοίγουν μια άλλη διάσταση. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο επίπεδο του συντονισμού ή επεξεργασίας ε, οδηγιών ή διαπιστώνοντας τις τάσεις στα κράτη-μέλη, ε, μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε αυτά τα πεδία. Συμφωνώ μαζί σας, είναι δραματική κατάσταση. Μια ολόκληρη γενιά μπορεί να χαθεί λόγω της ανεργίας των νέων. Ε, νέων που δεν ξεκινάνε μια καριέρα. Όσον αφορά την οδηγία απόσπασης των εργαζομένων, περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία την πρόταση. Δεν συμφωνούμε βέβαια με όλα τα σημεία που περιέχονται δεν θέλουμε να υπάρξουν ε, καταχρήσεις και να μεληθούν κάποιοι κλάδοι. Ίσως μπορούμε να πετύχουμε μια νομοθεσία αποτελεσματική που θα εντοπίζει και θα αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα όσον αφορά την απασχόληση. Χρειαζόμαστε μια νέα οδηγία όσον αφορά το θέμα. Όσον αφορά το Ταμείο για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, αυτό είναι ένα θέμα πιο προβληματικό. Μόνο το 1 τρίτο της οικονομικής πρικοδότησης που διατέθη χρησιμοποιήσαμε. Χρειάζονται νέες ιδέες. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης. Ζητούμε από την Δανική Προεδρία να προσέξει και αυτή την πτυχή. Όλα αυτά, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που αναφέρατε, όλες αυτές οι προσπάθειες που αναφέρατε, και στις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε θα είναι κάτι καλό. Και διακόπτει εδώ η πρόεδρος τον ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στις δύο υπουργούς και να ευχαριστήσω την Προεδρία βέβαια, εάν ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Έτος του 2012 για την ενεργή γύρενση και την ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ως εισηγητής λοιπόν θέλω να σας δω με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε αυτήν την αλληλεγγύη των γενεών και έχω και μια πρόταση η οποία έχει μεταβληθεί σε κοινή, σε γραπτή δήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς μπορεί να υπάρξει μια ε, δυνατότητα ε, αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών για να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο τους νέους αλλά και τους ηλικιωμένου. Να υπάρχει λοιπόν και μια συμμετοχή των ηλικιωμένων για την ε, αλληλεγγύη, την ενεργή μεταξύ των γενναίων και έχει σαν στόχο και την αξιοπρέπεια και την ζωτικότητα των γενεών και είναι πραγματικά σημαντικό να το υποστηρίξουμε γιατί αυτό έχει να κάνει και με την ζωτικότητα όλων των μελών της κοινωνίας ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Ελπίζω λοιπόν ότι με τα γεγονότα τα οποία θα διοργανώσετε και με τις προτάσεις σας θα μπορέσετε να προχωρήσετε τα θέματα αυτά σε αυτό το εξάμεινο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά τώρα για να διευκολύνω την κατάσταση, λέει η Πρόεδρος. Να θέσω δύο ζητήματα. Το πρώτο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι συζητήσεις για το πλαίσιο το νέο κανονισμό θα δεξαχθεί επί Προεδρία σας. Ελπίζω να μπορέσετε να σημειώσετε συγκεκριμένη πρόοδο στον τομέα. Στην παρούσα κατάσταση όμως αυτό που είναι κρίσιμο για μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να προσαρμοστεί αυτό στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Διότι ως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, δείχνει ότι είναι ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να αλλάξει επί να μετακινηθεί για πέντε χρόνια, όπου η αγορά εργασίας αλλάζει πολύ γρήγορα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε το Ταμείο πιο ευέλικτο και να είμαστε ευφυείς όσον αφορά την χρήση του εργαλείου αυτού. Γνωρίζω ότι δεν ισχύει αυτό τώρα. Αλλά αν πιστεύουμε ότι είναι εργαλείο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την οικονομική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό που προανέφερα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερη παρατήρηση. Την έκθεση για την ετήσια ανάπτυξη. Την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη. Θα θετήσουμε αργότερα την έκθεση τη κυρίας Κορνέλισεν, όπου σχολιάζουμε και έχουμε και προτάσεις τα όσα σχετικά με αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύουμε ότι αποτελεί πολύ καλή συνεισφορά αυτή για το Εαρινό Συμβούλιο. Θα ικανοποιούμε, θα λοιπόν τα μάλλον μπορούσε να σημειώσει και να λάβει υπόψη αυτή την έκθεση η Ιδανική Προεδρία και χρησιμοποιήσει την έκθεση σαν προστιθέμενη αξία για τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του Εαρινού Συμβουλίου. Βέβαια θα δώσουμε εντολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει αυτή τη θέση και να την πρασπιστεί στο Συμβούλιο Κορυφής. Αν θα μπορούσε με ανοιχτό πνεύμα να διαβάσει το κείμενο η Ιδανική Προεδρία θα ήταν πιο επικοδομητικό και θα βοηθούσε και εσά να τύχετε καλύτερη ισορροπία στις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Παρακαλώ λοιπόν να πάρετε τον λόγο τώρα για να δώσετε απαντήσεις και να προβείτε και στα τελικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για αυτή την έξοχη συζήτηση. Ναι, πραγματι, ως ε, Προεδρία ε, δεχόμαστε ευνοϊκά αυτή την έκθεση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη. Είναι μια υπόσχεση αυτή ότι θα τη λάβουμε υπόψη αυτή την έκθεση, μπορούμε να σας τη δώσουμε αυτή την υπόσχεση. Το μέλλον θα είναι σκοτεινό ή όχι. Νομίζω όχι. Ε, επί του παρόντος αντιμετωπίζουμε μια ευαίσθητη κατάσταση μέσα στην κρίση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η πρώτη φορά όμω, Αντιμετωπίσαμε και άλλε κρίσει κατά το παρελθόν. Αυτό που είναι σημαντικό και αποφασιστικό κατά την άποψή μα είναι η δυνατότητά μα ε, να στριμωχθούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε καινοτόμε λύσει ε, έναντι των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ξεκινώ αυτό το γύρο απαντήσεων υπογραμμίζοντας ότι πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει την οικονομική υπευθυνότητα με την πρόθεση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αυτό όμως απαιτεί να καθορίσουμε προτεραιότητες. Θα είναι ευαίσθητη η συζήτηση, δύσκολη συζήτηση που πρέπει να γίνει μεταξύ κρατών μελών. Το Ταμείο Προσαρμογής ε, στην παγκοσμιοποίηση είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Χρειάζεται πιο συγκεκριμένη συζήτηση βέβαια. Μετά μου θέσατε και άλλο ένα άλλο ερώτημα κατά πόσο μια νέα οδηγία απόσπασης ε, θα μπορούσε να ε, διατυπωθεί. Ξέρω ότι κάποιοι θέλουν μια τέτοια οδηγία, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε μια πλειοψηφία που θα ακολουθεί αυτή τη σχολή σκέψη. Και σαν χώρα που είναι στην Προεδρία προτιμούμε να παραμείνει η οδηγία και να εφαρμοστεί σωστά και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Ε, το οποίο είναι και αναγκαίο άλλωστε. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων εργαζομένων από τη μια και από την άλλη ε, αγορά εργασίας και κινητικότητα. Και εγώ εξίσου διερωτώ με κατά πόσο θα πρέπει να διοργανωθεί μια διάσκεψη ε, που θα αφορά το περιβάλλον εργασίας. Να το ετοιμάσουμε αυτό το, αυτή την εκδήλωση σαν Προεδρία. Είμαστε διαθέσιμοι να οργανώσουμε κάτι τέτοιο συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δει το φως της μέρας με τέτοια διάσκεψη, ούτω ώστε αυτή η νέα στατηγική για το περιβάλλον εργασίας για την περίοδο 2013-2020 ε, να δημιουργηθεί θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα, να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά έχω να καλύψω και άλλα δύο σημεία που ετέθησαν. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που υπόθηκε. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η εγκατάλειψη του σχολείου. Ε, είναι θετικό που αυτό αναφέρεται σαν προτεραιότητα στη Δυτική της Ευρώπης 2020. Είναι ένα στόχος τον οποίο επικροτώ ε, και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις εργασίες της Προεδρίας αυτό το θέμα. Αυτή η διάσκεψη θα οργανώσουμε εμείς τον Απρίλιο ε, στη Δανία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ακριβώς θα πρέπει να αναφέρεται σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας και τι σχέση έχουν αυτά με την ανεργία των νέων. Οι κοινωνικοί εταίροι ε, στη Δανία επανειλημμένα εξέφρασαν την επιθυμία να χρησιμοποιηθεί η παιδεία και η κατάρτιση. Και η θεωρία, η κατάρτιση και η εκπαίδευση να συνδυαστούν με την πρακτική εφαρμογή. Ε, νομίζω ότι εκεί εν μέρη έγκυται ε, ένα στοιχείο της λύσης που πρέπει να βρούμε. Διότι οι νέοι χρειάζονται ε, να μάθουν κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο και θα πρέπει να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Τέλος και κάτι συγκεκριμένο μου τέθη σε ερώτημα όσον αφορά την κατάσταση που ισχύει στην Πορτογαλία. Είναι ευαίσθητο θέμα, δεν σας το κρύβω. Ε, πρέπει να γίνουν απόλυσει ναι ου Να απολυθούν εργαζόμενοι. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η συζήτηση επί της αρχής. Αν θέλετε, αν προβλέπετε διευκόλυνση των απολύσεων από τη μία πλευρά, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που να είναι επαρκές. Και εδώ μιλώ προσωπικά. Ε, και εδώ μπαίνει και η ευελιξασφάλεια που προανέφερα. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση υψηλού επίπεδου που δεξήχθη και ελπίζω να σας δω ε, και στο μέλλον σε διάφορα άλλα βήματα. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Ε, είδατε σε ένα εξάμεινο σας ζητούμε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ευθύνη, έχει την ευθύνη της Προεδρίας μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι και ανησυχούν και έχουν και προσδοκίες. Περιμένουν μήνυμα από την Ευρώπη στον κοινωνικό τομέα. Λοιπόν, επομίζεστε τεράστιες ευθύνες. Τα μέλη της Επιτροπής είναι στο πλευρό σας όπως θα καταλάβετε, ούτως ώστε αυτό το εξάμεινο να είναι επιτυχές. Ραντεβού, λοιπόν, σε άλλες περιστάσεις κατά της Προεδρίας σας και ελπίζουμε η συζήτηση να είναι εξίσου πλούσια όπω η σημερινή και στο μέλλον. Καλή δουλειά, κάθε επιτυχία σα εύχομαι, εν ονόματι όλων των συναδέλφων τη Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ. Αν ναι, ναι, ναι, πείτε κάτι, μήπω. Λυπούμε, λέει Δηλαδή, Θέλω να σα ευχηθώ και να σα χειροκροτήσω. Νομίζω ξέχασα σε όσο το λόγο, αλλά έχετε δύο-τρία σημεία που θέλετε να αναφέρατε. Λοιπόν, ορίστε, πάρτε το λόγο. Ήθελα να, κάποια σχόλια να κάνω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, κυρία Μπερέ. Η Ευρώπη βασίζεται ε, πάνω μα να βρούμε λύσει. Να βρούμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σχόλια που ακούσαμε από εσά. Είπατε ότι ολόθερμα συμφωνείτε με το πρόγραμμά μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και ελπίζουμε σε μια μελλοντική καρποφόρα συνεργασία μαζί σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, επανέλθετε στις θέσεις σας. Στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης βρισκόμαστε τώρα και δίνω τον λόγο στην κυρία Κορνέλη Σεν που είναι η συγγήτριά μας για τα θέματα απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων για την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012 είναι ένα θέμα το οποίο θα έρθει στην Ολομέλεια μετά από την έγκρισή μας στην Επιτροπή μας και παράλληλα έχουμε τη γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ήδη εγκρίνει την έκθεση του κυρίου Γκοζέση σχετικά με τα θέματα αυτά. Κύριε Κορνέλσεν, μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις 25 τροπολογίες συνειβιβασμού που έχετε συντάξει μαζί με τους Σκιώδης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε μια πρώτη συζήτηση για το έγγραφο αυτό εργασία, επί τη, επί τη βάση αυτού του εγγράφου. Φυσικά θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το έγγραφο εργασία για να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής. Ένα από τα κύρια μηνύματα των άλλων πολιτικών ομάδων από την αριστερά μέχρι τη δεξιά στη συζήτηση αυτή είναι ότι η ανεργία των νέων είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, στην έκθεση η οποία έχει προέλθει από αυτή τη συζήτηση, έχω προσθέσει και το θέμα της αντιμετώπιση, της ανεργία των νέων σε ένα από τα κέρια μηνύματά μας. Σχεδόν όλες οι τροπολογίε οι οποίες έχουν υποβληθεί είναι ιδιαίτερα θετικές και πολύτιμέ προσθήκες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για το γεγονός ότι μπορέσαμε να συντάξουμε περιεκτικές συμβιβαστικές λύσεις. Σχεδόν τελείωσαν τα γράμματα του αλφαβήτου για να τις ονοματίσουμε. Ελπίζω λοιπόν <clears throat> ότι θα μπορέσουν να συλλέξουν μια ευρεία πλειοψηφία και εδώ και στην Ολομέλη αυτές οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Εγώ λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ με το να υπάρξει και κάποια μεγαλύτερη προσοχή από το Συμβούλιο για τις προσπάθειές μας και θέλω να ευχαριστήσω και την ε, Πρόεδρο για το σαφές μήνυμα που έδωσε στις δύο Υπουργούς προηγουμένως σε στενή συνεργασία με τον κύριο Γκοζές, ο οποίος είναι ο εισηγητής στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, όπως είπα. Θα συναντηθώ με, και με τον πρόεδρο τον κύριο Σούλτς και με την Προεδρία της Κομισιόν, ώστε να μπορέσουν να γίνουν σαφείς οι προτεραιότητές μας και να έρθουν στην πλήρη γνώση τους. Θα ήθελα να ζητήσω από τους σκιώδεις συζητητές και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, εάν θέλουν να κάνουν κάποια περαιτέρω συμβολή ε, και αν μπορούν να συζητήσουν και με τους μόνιμους εκπροσώπους τους στην Κορεπέρ για να μπορέσει να προωθηθεί το θέμα αυτό. Όλα αυτά θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και αν οι, βασικέ οι βασικές μας προτεραιότητες γίνουν δεκτές από το Συμβούλιο, όχι μονάχα θα διασώσουμε το ευρώ, αλλά θα διασώσουμε και τους πολίτες. Θα συνεργαστούμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κορνέλσεν. Μπορεί να είναι ε, υπερήφανη για την έκθεση αυτή και αυτό το οποίο λέτε ότι πρέπει να σώσουμε όχι μόνο το ευρώ αλλά και τους πολίτες μας είναι πολύ σωστό. Πρέπει να γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες, όλα τα δυνατά διαβήματα προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και την Δανική Προεδρία για να ληφθούν υπόψη οι θέσεις μας για τα ζητήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Κονέλσεν για το έργο της, την ευκαμψία που έδειξε. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με τις τροπολογίες αυτές. Εγώ θα υποστήριζα το L και την τροπολογία S λατινικό όταν μιλάνε για ίση αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις αποδοχές και το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο Πέραν αυτού έχω να κάνω μερικά σχόλια πολύ σύντομα για ορισμένε τροπολογίε. Εμείς θέλουμε να ζητήσουμε μία χωριστή ψηφοφορία στην τροπολογία 83 για την ε, χωριστή σύσταση ε, για τη χωριστή μάλλον καταγραφή συστατικών στοιχείων για τους νέους και επίσης για την 114 θέλουμε πάλι μια χωριστή ψηφοφορία και στη 47 σε σχέση με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω κυρία Κονέτσα για την πολύ καλή σας έκθεση. Ίσως τα έχω μπερδέψει λέει η πρόεδρος. Αναφέρεστε σε τροπολογίες που έχουν αριθμούς, όχι γράμματα. Δεν είναι μέσα στις τροπολογίες συμβιβασμού. Κατάλαβα λάθος. 47, όχι 7 λέει η κυρία Χάρκιν. Κυρία Γιαζοβιεύσκα. E, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι έξοχο το έγγραφο αυτό. Αυτή η τύση ανάλυση εν γέννη είναι ένα είδος δοκιμής, τεστ που κάνει μια αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλά και των προγραμμάτων των κρατών μελών σε αφορά την κοινωνική πολιτική, την πολιτική απασχόληση. Να σε πιστήσω την προσοχή επί κάποιων τροπολογιών που κατέθεσα που θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, ανάλυση της ανάπτυξης αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν την απασχόληση σε κάθε νέο, αν τεθεί αυτός σαν στόχος, είναι στόχος ανέφικτος. Ε, θα πρέπει να λέμε ότι θα δίνεται δυνατότητα στους νέους, παρέχεται υποστήριξη στους νέους όσον αφορά το επιχειρήν. Και σαν στόχος θα πρέπει να παραμείνει η βελτίωση του συστήματος του εκπαιδευτικού, ώστε οι δεξιότητες που αποκτώνται στο σχολείο να αντιστοιχούν στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Δεύτερον, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική δραστηριότητα πιο βιώσιμη. Αυτό είναι κάτι που υπογραμμίζεται στο έγγραφο της εισηγήτριας και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να άρουν τους φραγμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν και που δυσκολεύουν την ανταλλαγή εργατικών χεριών μεταξύ ε, κρατών μελών. Και έτσι δεν μπορεί να γίνει πλήρης χρήση των ανθρωπίνων πόρων ε, στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Ε, ακούγοντας τις δύο κυρίες υπουργούς, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αυτές οι προτεραιότητες. Νομίζω ότι υπογραμμίζει σωστά αυτές τις πτυχές το έγγραφο. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κ. Γιάννος Σλόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ως ε, σκιώδης ε, εισηγητής για την έκθεση της κυρίας Κορνέλισεν. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, που ασχολήθηκε με αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Κορνέλισεν για την τέλεια συνεργασία μας και κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα διότι πίεζε ο χρόνος. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Καταφέρατε κυρίες ηγήτρια να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες μας όλες και τα αιτήματά μας. Είναι τέλεια η έκθεση και αναφέρεται σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα προγνωστικά για το 2012, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η πιθανότητα... το επίπεδο της ανεργίας θα παραμείνει πάντα πολύ υψηλό. Αυτό που με εκπλήσει στο πλαίσιο αυτό είναι ότι από το 2009 ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δεν καλύπτονται αυξάνεται επίσης. Άρα θα πρέπει πραγματικά να βασιστούμε σε ένα καλό σύστημα κατάρτισης και να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ε, θα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, από το δημοτικό μέχρι τις ε, σπουδές τις πανεπιστημιακές. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, μαθητεία, να βελτιώσουμε την κινητικότητα να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Τα ευρωπαϊκά εργαλεία είναι πολύτιμα. Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να συνδέσουμε με δράσεις πρόθεσης της οικονομικής ανάπτυξης και με την πολιτική απασχόλησης. Είπατε ότι η νεολαία πλήττεται περισσότερο από αυτή την κρίση. Την περίοδο 2008 με 2010 συνολικός αριθμός ανέργων κάτω των 25 ετών αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο άτομα ένα εκατομμύριο άτομα παραπάνω. 40% των νέων εργάζονται, μάλλον δεν εργάζονται και δεν έχουν τη δυνατότητα ε, να βρουν κάποια εργασία διαρκείας. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αύξηση των ευκαιριών που δίνονται στους νέους πιστεύω ότι θα ε, μας βοηθήσει να κινηθούμε σωστά για να αντιμετωπίσουμε το, την ανεργία. Ε, ε, ε, θα μπορούσαμε μέσω των προγραμμάτων έρευνας να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις για να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ο κύριος Πέκερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Και εγώ. Ευχαριστώ για την εργασία αυτή, διότι η συγκεκριτής κατάφερε να συγκεντρώσει, να συνδυάσει συγκεκριμένα στοιχεία και να τα συνθέσει. Η τελευταία τροπολογία που αναφέρατε μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική γιατί ζητάει από τα κράτη-μέλη και τις εθνικές κυβερνήσεις να αντιδράσουν άμεσα και αποφασιστικά και να εφαρμόσουν αυτά που και τα ίδια αποφάσισαν στο Συμβούλιο δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι συμφωνίες αυτές, οι αποφάσεις αυτές του Συμφουλίου δεν εφαρμόζονται αφού πρόκειται για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αξιοδότησης, αγοράς εργασίας, γιατί δεν εφαρμόζονται. Δεν μπορούμε να λέμε δεχόμαστε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την ενεργό γύρανση αν δεν υπάρξουν σχετικές μεταρρυθμίσεις και αν οι μεταρρυθμίσεις που συστήνονται δεν εφαρμόζονται. Το χρωστάμε αυτό στις επόμενες γενιές νομίζω. Αλλιώς δεν θα μας πιστεύουν πια, δεν θα πιστεύουν καμία μας υπόσχεση οι νέοι, ούτε οι γυρεότεροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για το πνεύμα με το οποίο συνέταξε την έκθεσή της που είναι τόσο ρεαλιστική και που λαμβάνει τόσο καλά υπόψη της και τα πραγματικά στοιχεία και τις συζητήσει του Συμβουλίου της Μακροοικονομικές γενικότερα. Νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει έτσι στην Δανική Προεδρία είναι σημαντικό παραμένει να το συνεχίσουμε, να χρησιμοποιούμε και εμείς την ίδια προσπάθεια. Έχω όμως μία πρόταση. Την είχα αναφέρει και στη συνάντηση των σκιωδών και από τότε δεν το είχα υποβάλει γραπτός, με συγχωρείτε. Μια προφορική λοιπόν τροπολογία που να αναφέρει τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ως προς την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανέχειας. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό ως μία παύλα του σκεπτικού για να αυξηθεί έτσι λίγο η δυναμική της έκθεσης. Ελπίζω να μην υπάρξουν αντιρρήσεις. Θα κάνω σχετική πρόταση γραπτό το απόγευμα, αλλά με ως προφορική τροπολογία. Σύμφωνα με, τις με τα τελευταία στοιχεία του Eurostat, το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι αναμένουν από εμά κατά προτεραιότητα πώς θα καταπολεμήσουμε την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο. Θα δώσω λοιπόν ξανά το λόγο στην εισηγή του Ρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν εδώ στη συζήτηση. Δεν θα επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες που τέθηκαν. Ε, πάντοτε θα υπάρχουν διαφορές για τις μικρολεπτομέρειες μεταξύ ομάδων. Αλλά γενικά νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και θα υπάρξει μεγάλη συνένεση. Και στην Ολομέλεια ελπίζω να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία για να μπορέσουμε να πούμε ιδού η εντολή που δίνουμε στον κύριο Σούλτς. Αυτό είναι η άποψη σχεδόν του συνόλου του Κοινοβουλίου δηλαδή. Θα προσπαθήσω να πείσω και την κυρία Χάουγκ για το συνδυασμένα στοιχεία που ρώτησε, που ζήτησε και φυσικά δέχομαι την προσθήκη μιας παύλας για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμηση της ανέχειας. Έτσι ενδυναμώνεται το κείμενο. Αυτά λοιπόν σας ευχαριστώ και προσμένω την ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο και θα πάει στην Ολομέλεια στις 15 Φεβρουαρίου σε κοινή συζήτηση μαζί με την έκθεση Γκονζές. Καλά είναι για αρχή του χρόνου. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 11. Προηγουμένως όμως θέλω να ξέρετε, να ξέρουν οι συντονιστές και συντονίστριες καθώς και οι υπάλληλοι των ομάδων ότι το σημείο που προσθέσαμε στην ημερήσια διάταξη στο τέλος τη αιτήση του συντονιστή του ΕΛΚ, δηλαδή τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί αύριο για την ψηφοφορία επί του, 28, επί του 27, θα γίνει και κλεισμένον των θυρών για προφανείς λόγους. Το 11 λοιπόν τροποποίηση του κανονισμού για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλεια και του κανονισμού και καθορισμό τη διαδικασία εφαρμογή του κανονισμού. Ο κύριο Κάμπρνοχ για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδης, σε εσά απευθύνομαι καταρχάς για να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που είχαν την καλοσύνη να υποβάλουν τροπολογίας. Με διορία την 11η Ιανουαρίου. 25 τροπολογίες κατατέθηκαν, ορισμένες μαζί άλλες μία-μία και 8 ακόμη άλλες εξετάζονται. Είμαι πεπισμένος ότι αυτοί που τις υπέβαλαν, αυτοί που τις συνέταξαν θα τις υποβάλουν κατά τη συζήτηση που θα ακολουθήσει ο κανονισμός για την αλλαγή του οποίου συζητούμε νομίζω ότι συμβαδίζει Δεν θα θέσει προβλήματα και στους εθνικούς νομοθέτες, αν και είναι σοβαρά και πολλαπλά τα προβλήματα των κοινωνικών δαπανών που πρέπει να συμφωνούν με τον, κάθε προϋπολογισμό, τον της κάθε χώρας. Είναι υποχρεωτικό αυτό, υποχρέωση του εθνικού προϋπολογισμού. Θα ήθελα να πω γενικά ότι οι τροπολογίες αφορούν κυρίως τρία θέματα. μεταξύ των οποίων την επίσημη έδρα και τις αποζημιώσεις για τους ανεξάρτητους διαμεθοριακούς. Σκοπός μου είναι να εγκριθεί από την πρώτη ανάγνωση και γι' αυτό θα ήθελα ήδη να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα προηγουμένως, όταν συζητήθηκε αυτή η έκθεση την πρώτη φορά. Οι περισσότερε τροπολογίες έχουν τεχνικό χαρακτήρα και οι συμβιβαστικέ τροπολογίες βέβαια και αυτές εξ ανάγκη έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Για ορισμένε τροπολογίες και για τη διατύπωσή τους, για την 15, 16, 17, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, διατύπωσή τους από ότι η 18. Και επίσης η 26 έχει καλύτερη διατύπωση από την 27 για τους κοινωνικούς εταίρους. Το να προσθέτουμε τη διατύπωση κοινωνική εταίρη στο κείμενο αυτό δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη σαφήνεια. Και όπως είπε και ο εισηγητής, προηγουμένως. Είναι σημαντικό για μας να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τη γραμμή που ενέκρινε το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη μεταφορά ε, επιδομάτων ανεργίας. Ελπίζω μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για το θέμα αυτό. Κύριε Θέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κλαπνόχ και το πνεύμα διαλόγου και συνεργασίες που είχαμε μαζί του ως σκιώδεις συγητές και να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και την προσπάθεια και του Συμβουλίου για να μπορέσει να καταλήξει σε μια συμφωνία που μας φαίνεται όλους να είναι λογική παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες που είχαμε για αυτή τη συμφωνία. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν όλες τις τροπολογίες των σοσιαλιστών γιατί θεωρούμε ότι βελτιώνουν το κείμενο και εάν απαραίτητο θα αποσύρουμε κάποιες από αυτές για να επιτευχθεί μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Είναι σημαντικό να δοθεί η νομική ασφάλεια, η ασφάλεια δικαίου στους εργαζομένους οι οποίοι είναι διακινούμενοι μέσα στην Ευρώπη γιατί η εξασφάλιση των κοινωνικών τους παροχών δίνει νέα δικαιώματα στους εργαζομένους Ιδίω σε αυτούς οι οποίοι γίνονται άνεργοι και ιδίω θεσπίζει ένα προηγούμενο σε σχέση με τις αποδοχές τους και τις επιβαρύνσεις που στις οποίες και με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναχαιτήσει την προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων που μετακινούνται με δόλιους σκοπούς και για να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος τους. Πρέπει εδώ να υπάρξει και η απαραίτητη παρακολούθηση για να δούμε αν στην πράξη αυτό το νομοθέτημα οδηγεί σε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση και έχει ο κ. Κράχνο την υποστήριξη των σοσιαλιστών. Η κυρία Οβίερ. Ε, Κυρία Πρόεδρε. Laudadele Αυτός ο κανονισμός έρχεται ενώπιόν μας επειδή το 2009 δεν είχαν καλυφθεί στην τροποποίηση του προηγούμενου κανονισμού ορισμένοι τομείς που ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων επί 10 χρόνια και παραπάνω. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης έχουν τροποποιηθεί σε πολλά κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ <clears throat> δεν είναι πάντα επίκαιρα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο κανονισμός να αντιμετωπιστεί από όλους με τον ίδιο τρόπο. Εγώ ως εκπρόσωπος των φιλελευθέρων πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες είχαν σαν σημείο ε, εκκίνησης να διασαφηνίσουν καλύτερα τον κανονισμό αυτό. Είναι πολλές ε, τροπολογίες οι οποίες είναι παρόμοιες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε επιτύχει το στόχο αυτό. Συμφωνώ <clears throat> με τον εισηγητή. και είναι δική μου, και δική μου επιθυμία να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση αυτό το νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Καταρχώς ευχαριστήσω τον κ. Καμπορ γιατί είναι πολύ λεπτομερής και στατηγική η δουλειά που έγινε όσον αφορά το κείμενο. Εν γέννη, αυτή η τακτική αναθεώρηση ε, έχει σημασία να μην διαλύει αυτό που οικοδομήσαμε επί σειρά ετών. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Στα πλαίσια του business friendly να προσαρμόζουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στις επιθυμίες των επιχειρήσεων περισσότερο από ότι για την αντιμετώπιση ε, της κατάστασης που και του εργαζομένους. Επανειλημμένα συζητούμε το πώς εξασφαλίζουμε την κοινωνική προστασία και την ισότητα των δικαιωμάτων εκείνων που τελούν υποκινητικότητα και να μην δημιουργήσουμε μια κατάσταση που ευνοεί ένα κοινωνικό ντάμπινγκ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εξέταση του θέματος του προσωπικού αεροπορικών εταιριών κυρίως. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με το θέμα, τον κύριο Τάγκερ. Θέλουμε τεχνική άποψη. Την αξιολόγησή σας σε συνάντηση με συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο και τις προτάσεις που γίνονται. Ευχαριστώ πρόεδρα, Όπως ήδη εξήγησα, σε πρώτερη συνάντησή μας, είναι τακτικό το εγχείρημα αυτό της ε, ενημέρωσης του κανονισμού για την κοινωνική ασφάλιση. Όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται επικαιροποίηση των νέων κανονισμών που ετέθησαν σε ισχύ μόλις την 1η Μαΐου του 2010 μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεις. Στις προηγούμενες, σε προηγούμενες κανονισμούς γινόταν επικαιροποίηση τεχνικού χαρακτήρα ετησίως. όπως σωστά σημειώθηκε από κάποιες παρεμβάσεις, στόχος της ενημέρωσης του κειμένου να λάβουμε υπόψη την αλλαγή νομοθεσιών στα κράτη-μέλη. Αλλαγές που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη των πραγματεύσεων για τον νέο κανονισμό μέχρι ότου υποβληθεί πρόταση για τις αλλαγές αυτές και διορθώθηκαν και κάποια σφάλματα όσον αφορά το κείμενο των νέων κανονισμών. Και χρειάστηκαν και κάποιες διευκρινήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη το επτάμενο προσωπικό, το περίφημο. Και θέλαμε να καλύψουμε κάποια κενά για πολύ λίγους όπως τα επιδόματα ανεργίας για κάποιους αυταποσχολούμενους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Από τη σειρά μας, από την πλευρά μας μάλλον, καλωσορίζουμε τα όσα είπε ο εισηγητής, ότι θέλει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Τον ευχαριστούμε για τη θετική και επικοδομητική παρέμβαση που έκανε σε αυτή την Επιτροπή. Μη λησμονούμε ότι σε μια μια πρώτη τροποποίηση αυτών των τροπολογιών όχι μόνο θα αφελήσει τους διάφορους φορείς κοινωνικής πρόνοιας που θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς και που χρειάζονται διευκρινήσεις για να εφαρμόσουν σωστά τους κανονισμούς, βοηθά και αυτούς, αλλά είναι κάτι υποφελές και για τους πολίτες. Ακούσαμε δύο παραδείγματα. Δηλαδή ποια είναι εφαρμοστέα νομοθεσία για το επτάμενο προσωπικό των εμπορικών εταιριών και κάλυψη κάποιων αυτοποπασχολούμενων μεθοριακών εργαζομένων. Και είναι καλό που υπόθηκε ότι υπάρχει επιθυμία να πετύχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, θέλετε να ολοκληρώσετε αυτή τη συζήτηση, να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο και όλους όσους μέσω θετικής προσέγγισης επέτρεψαν να ετοιμάσουμε αυτή την έκθεση και να προετοιμάσουμε αυτή τη νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Όσον αφορά αυτό το θέμα λοιπόν και από αυτής της θα πω ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση στις 29 Φεβρουαρίου. Άρα έχετε χρόνο για να επεξεργαστείτε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Και θέλουμε, όπως είπατε, θέλετε η υιοθέτηση ε, του κειμένου σε πρώτη ανάγνωση. Πάμε στο σημείο 12 της ημερήσιας ε, διάταξης. Η συγγετής είναι ο κ. Τσάμπα Ορή. Εξετάζεται όλο το πακέτο της απαλλαγής του προϋπολογισμού του 2010 αφορά το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενική απαλλαγή όσον αφορά την επίδοση την οικονομική και τον έλεγχο των υπηρεσιών της Ένωσης, το Ίδρυμα για την κατάρτιση, δηλαδή τα Ιδρύματα Κατάρτισης, το Ίδρυμα του Τωρίνου, το Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων εργασίας, δηλαδή του Δουβλίνου, το Ίδρυμα για την βετίωση ε, της Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ε, κύριε Σιγητά, σας δίνω το λόγο. Σχιώδες εισηγητές είναι οι ίδιοι για όλο το πακέτο, άρα σας προτείνω να μας παρουσιάσετε γενικά την απαλλαγή επί των έξι κειμένων και μετά θα διεξαχθεί η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας. Αλλά εάν δεν είχατε προτείνει εσείς να το δούμε αυτό το θέμα ως θέσμη, όλες αυτές τις απαλλαγές, θα το είχα προτείνει ίδιο ο ίδιος. Έρχομαι από το, το τέλος σε ό,τι αφορά την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, που είναι η βάση της εργασίας μου, πρέπει να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που μπόρεσα να κάνω μια πρόταση η οποία περιλαμβάνει απλώς τη διαπίστωση ότι οι αποκεντρωμένοι φορείς έχουν εργαστεί με τρόπο νομότυπο και απόλυτα σαφή σε επίπεδο δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό το οποίο λέει το ελεκτικό συνέδριο είναι ότι έχουν εργαστεί με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί οι αποκεντρωμένοι φορείς. Είναι μια ευκαιρία για μένα να συγχαρώ τους αποκεντρωμένους φορείς. Υπήρξε στο παρελθόν εισηγητή για τα θέματα αυτά και στα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πάντα σημεία που έδιναν λαβή σε κριτικέ και είχαμε πάντα ζητήσει από του φορείς αυτού να διορθώσουν κάποια πράγματα. Εφέτο δεν ισχύει κάτι τέτοιο και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητώ την απαλλαγή όλων αυτών των φορέων. Θέλω να ευχαριστήσω και το ελεκτικό συνέδριο. Είναι απόλυτα εντάξει η προπολογισμή και η εκτίμηση, η εκτέλεση των προπολογισμών αυτών των φορέων και αυτό είναι ακριβώς και αυτό στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η επί ε, Επιτροπή. Θα ήθελα τώρα να κάνω και κάποια σχόλια για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή. Εδώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μόνο 18% από τις δαπάνες της ε, πολιτικής συνοχής αφορά τον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών έχουν το 95% έχουν καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θετικό λοιπόν το να δούμε ότι το 80% σε πιστώσεις πληρωμών και το 100% των πιστώσεων υποχρεώσεων έχουν πράγματι το 100% των πιστώσεων υποχρεώσεων έχουν ε, πράγματι δεσμευτεί. Είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό στις ε, πιστώσεις πληρωμών. Εδώ πρέπει να υπάρξουν λοιπόν βελτιώσεις στον τομέα του Ταμείου Συνοχής, ιδίως ε, στη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης οικονομικής. Και υπήρξαν και προβλήματα μεμονωμένα σε συγκεκριμένα σχέδια και εδώ το πρόβλημα είναι ότι η σύνεψη υποχρέωσεων έγινε πολύ καθυστερημένα, επομένως δεν μπορούν να εκταμιευθούν οι πιστώσεις πληρωμών και στον ίδιο χρόνο που γίνεται η δέσμευσή τους. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να υπάρξει προσπάθεια να γίνεται το ταχύτερο, να γίνεται πιο πρόημα η δέσμευση υποχρεώσεων, ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα τα χρηματοδοτικά και να μην χάνονται στο τέλος του χρόνου. το ποσοστό των σφαλμάτων και των ατελειών ήταν πολύ χαμηλό, 7,7%. Εδώ μπορεί ο καθένας να έχει διαφορετική άποψη αν είναι πολύ χαμηλό ή πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό. Και υπήρξε και κάποια δυσκολία στον ορθό προσδιορισμό του ποσοστού αυτού σφαλμάτων στην, ε, στην ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είναι σίγουρο ότι έχει μειωθεί το ποσοστό των σφαλμάτων και αυτό είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, την οποία εγώ χαιρετίζω. Χαιρετίζω περαιτέρω και το γεγονός ότι η Κομισιόν προσπαθεί να συρρυκνώσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό αυτών σφαλμάτων με την παροχή συμβουλών, με καλύτερη εκπαίδευση, με διαβουλεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Επομένως και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικροτήσουμε αυτές τις θετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν και σύμφωνα επίση και με την παρατήρηση που έγινε ότι τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, κονδυλίων αυτών θα πρέπει να τηρούν την υποχρέωση του να δίνουν εκθέσεις στην Κομισιόν και η Κομισιόν αντιστοίχω να προβαίνει στην αξιολόγηση και τον έλεγχο αυτών των εκθέσεων ώστε να διασφαλίζει ότι οι απαραίτητες πληρωμές έχουν καταβληθεί πλήρως. Και είναι σύνομες. Είπα προηγουμένως ότι όπως και στο παρελθόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια στενή συνεργασία με την Όλαφ, με το γραφείο λοιπόν για την καταπολέμηση της απάτης, γιατί αυτό θα μπορέσει να αποτρέψει τη δημιουργία προβλημάτων ή να επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωσή τους. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και από τα κράτη-μέλη στο τομεί των αρμοδιοτήτων να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να υπάρξει πιο στεναρή αντιμετώπιση των απατών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δίνουν και πιο ενδελεχείς εκθέσεις και αυτό θα δίνει καλύτερη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική κατανομή και χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Υπήρξαν σε ορισμένε περιπτώσεις προβλήματα που δεν ήμασταν σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε, παραδείγματος χάρη στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας. Και έχω πει στην ε, κυρία Υπουργό, ότι μόνο το 1 τέταρτο των κονδυλίων έχει χρησιμοποιηθεί και ίσως αυτό είναι ένας λόγος να περιοριστούν τα κονδύλια. Αν προτείνει η Κομισιόν να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη των κονδυλίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε με αυτό. Αλλά το στόχο μα θα πρέπει να είναι πάντα να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να εκταμιεύονται πλήρω. Θα πρέπει επομένω και η Κομισιόν να προσπαθήσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά, ώστε να είναι πιο σωστά τα σχέδια, μεγαλύτερη ποιότητα τα σχέδια τα οποία προτείνουν στα πλαίσια του ταμείου αυτού, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα υποστήριξη αυτών των κονδυλίων. Ίσως είναι πολύ, πολύπλοκες οι διαδικασίες και δεν είναι αρκετά γνωστές στους ε, υποψηφίους ε, να υποβάλουν σχέδια αυτές τις προδιαγραφές. Αλλά από τη δική μας πλευρά το απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει απώλεια αυτών των κονδυλίων, ότι τα κονδύλια αυτά τα οποία θα έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, ιδίως όταν χάσουν τη θέση εργασίας τους, πράγματι να υποφολούνται από αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν πολλέ ανάγκε λοιπόν, το εξασφαλίσουμε αυτό και με καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των υπευθύνων. Και πιστεύω ότι και από το σχέδιο του, από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι χρήσιμο να ξέρουμε και πώς προχωρούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες για την τόνωση της απασχόλησης, κάτι το οποίο θα διαλύσει και την δυσπιστία που υπάρχει πολλές φορές σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό μπορούμε να έχουμε και εδώ μια θετική αντιμετώπιση όπως τελείως θετική ήταν και η στάση μου εναντί των αποκεντρωμένων φορέων που είπα προηγουμένως ότι έπραξαν τα πάντα αγαστά και σωστά και αυτό θα ενισχύσει την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς φορείς. Και πάλι έρχομαι σε μια γενική παρατήρηση. Είπα ότι συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία διαπιστώνει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά πρέπει εδώ να κάνω μια μικρή μοναχά παρατήρηση. Νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα λυσιτελές να υπάρχει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αποκεντρωμένων φορέων μια καλύτερη συνεργασία. Αυτό θα μπορούσε να γίνεται παραδείγματος χάρη μέσα στα πλαίσια της εξέτασης του ετησίου προγράμματος εργασιών είναι όμως απαραίτητη να γίνεται πάντα μια προσαρμογή σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον. Επίσης να υπάρχει καλύτερη συνεργασία για τα θέματα του διορισμού των διευθυντών των αποκεντρωμένων φορέων. Κατακλείδει όλες αυτές οι σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τους αποκεντρωμένους φορείς να γίνονται με στενότερη συνεργασία και διαβούλευση και με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Ελέγχου του και την Επιτροπή Απασχόλησης. Ένα πρόσθετο σημείο το οποίο τόνισα στην πρότασή μου είναι ότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι αποκεντρωμένοι φορείς το ίδιο καθεστώς. Δεν θέλω τώρα να μπω στις λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να διατυπωθεί αυτό το ενιαίο καθεστώς, απλώς θέλω να πω ότι θα ήταν πραγματικά ε, αξιέπαινο και πολύ χρήσιμο να υπάρχει το ίδιο καθεστώς σε όλους τους αποκεντρωμένους φορείς. Και πιστεύω ότι σε όλους τους φορείς, όχι μόνο τον φορέα του Τωρίνο, να υπάρχουν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, αλλά σε όλους τους αποκεντρωμένους φορείς να υπάρχουν εκπρόσωποι που έχουν διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα μπορούσε επομένως να εξασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Να είναι χρήσιμο λοιπόν να υπάρχουν εκπρόσωποι οι οποίοι πράγματι θα συμμετέχουν ενεργά στα διοικητικά συμβούλια αυτών των φορέων. Επίσης, είχε προτείνει στον τομέα αυτό και το ελεκτικό συνέδριο να κάνουμε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κατάρτιση του προϋπολογισμού σε σχέση με την διάκριση, τη σαφέστερη διάκριση μεταξύ ε, δαπανών για προσωπικό και λειτουργικών δαπανών. Αν μπορέσει αυτό να επιληθεί το πρόβλημα, τότε μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερη συνεργασία με τους αποκεντρωμένους φορείς. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να γίνει και μία ενδελεχέστερη έκθεση για τη λειτουργία των φορέων σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές και τους κανόνες λειτουργίας τους, χωρίς όμως αυτό να συμφισβητείται η ορθότητα των ενεργειών τους. Μπορώ και πάλι, όπως είπα και προηγουμένως, να πω ότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εμά, όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους διοικητικούς τομείς να προβούν σε εξοικονομήσεις. Υπάρχει η αρχή αυτή της λιτότητος, η οποία θα πρέπει να ισχύει για όλους τους τομείς, για όλα τα θεσμικά όργανα και τους αποκεντρωμένους φορείς. Επομένως και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το ελέγχουμε και στο μέλλον. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούν να προκύψουν περαιτέρω εξοικονομήσεις και ίσως τα χρήματα τα οποία εξοικονομούνται θα πρέπει να απελευθερωθούν για σχέδια τα οποία θα είναι υποφελή. Αυτές ήταν λοιπόν οι παρατηρήσεις μου και οι προτάσεις μου και μπορώ να σας επαναλάβω ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να συγχαρούμε όλους τους αποκεντρωμένους φορείς και να αναγνωρίσουμε την σωστή της εργασία. Το απόγευμα θα έχουμε τους εκπροσώπους ορισμένων αποκεντρωμένων φορέων και μετά από πολλά χρόνια αποστόνισε προηγουμένως είναι η πρώτη φορά που στη διαδικασία της απαλλαγής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προτείνω επομένω να εγκρίνουμε την απαλλαγή αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κάνετε κάποια σχόλια όσον αφορά τους ε, οργανισμούς αποκεντρωμένους. Θα μπορείτε να τα ξαναπεί το απόγευμα θα είναι εδώ εκπρόσωποι του και θα διεξαχθεί μια ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Η κυρία Λάμπερτ. Έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την καθυστερημένη άφηξη. Για μερικές από αυτές τις εκθέσεις θέλουμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Όλα αυτά βέβαια θα ξανασυζητηθούν στην ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου με, για τη συνεννόηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Υπάρχουν ορισμένα θέματα για την εκπροσώπηση ιδίως. Τέλος πάντων τα βλέπουμε αυτά, τα βλέπουμε και στις ετήσιες εκθέσεις και κατά την παρουσίαση των ε, προϋπολογισμών των διαφόρων οργάνων. Ο συντονισμός και η απλοποίηση μεταξύ των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο επανειλημμένως έχουμε ζητήσει και βλέπουμε ότι χρειάζεται παραπάνω ή μάλλον έχει γίνει μια προσπάθεια να εφαρμοστεί, κάποια παραπάνω προσπάθεια. Το θέμα της εκπροσώπησης του Κοινοβουλίου στην ομάδα εργασίας αυτήν έχει γίνει θέμα συζήτησης πολλές φορές. Και στα συμπεράσματα όπου υπάρχει διαμάχη από αυτού με το, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θέλουμε να το βάλουμε γιατί η εκπροσώπηση αυτή του Κοινοβουλίου διαφέρει σε μερι, Μερικές φορές έχουμε πολλούς άλλες λίγους και δεν χρησιμοποιούμε όλη την ίδια γλώσσα. Η ομάδα μου λοιπόν θα εξετάσει την περίπτωση να υποκαταθέσει ορισμένες τροπολογίες οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν αναγκαστικά υψηλό κόστος λειτουργίας, όχι αναγκαστικά λέω εξαρτάται από το μέγεθός των. Όσο για το outsourcing και τον συνδυασμό υπηρεσιών πρέπει να ξέρουμε από ποιον προϋπολογισμό προέρχονται αυτά. η διαχείριση του προσωπικού και αυτή μπορεί να έχει ορισμένα προβλήματα ως προς τις μικρότερες ιδίως, τους μικρότερους οργανισμούς αυτούς. Και θέλουμε επίσης να επιμείνουμε στην έννοια του activity-based budgeting που λέμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά σχολιάκια, τρία δηλαδή. Πρώτον, υποστηρίζουμε τον εισηγητή για την απαλλαγή των υπηρεσιών. Τον συγχαίρω και εγώ, όπως συγχαίρω και τις υπηρεσίες για τη δουλειά τους που όπως έκανε και εκείνο. Τώρα για το τμήμα τρία κομισιών, γενικά γενικά, βασικά, συμφωνούμε, αλλά παρόλα αυτά θα καταθέσουμε τροπολογίες. Όπως για την παράγραφο 10 για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συμφωνούμε μεν, αλλά θα βάλουμε κάποιους καινούριου χρωματισμούς για να είναι τα πράγματα σαφέστερα. Για την παράγραφο 11 Επίσης θα καταφέρσουμε τροπολογία λέγοντας ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί σαφέστερα το κοινωνικό ταμείο από το περιφερειακό του. Καλό είναι να αποσεφινιστεί και αυτό. Τρίτον, για την τελευταία έκθεση Εκεί θα καταθέσουμε επίσης μερικές τροπολογίες για να αποσαφηνίσουμε πάλι ορισμένες παραγράφους τεχνικά. Ειδικότερα την 2 και 4 με τον ορισμό του διευθυντού, τον υπηρεσιακό κανονισμό και υπαλληλικό κανονισμό κλπ. Να, αυτά είναι το που θα καταθέσουμε. Γενικά όμως συμφωνούμε με τον εισηγητή και σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κανεί άλλο, καμία άλλη. Όχι, επομένω ο εισηγητή. Ευχαριστώ. Περιμένω λοιπόν με περιέργεια να δω τις τροπολογίες και τις προτάσεις των συναδέλφων και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω αυτές τις προτάσεις. Κατά την άποψή μου, με καλή διάθεση μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα καλό κείμενο. Γιατί όχι λοιπόν. Τώρα δεν είδα πώς μπορούμε στις διάφορους επικεντρωμένους οργανισμούς να εκπροσωπηθούμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε μία αρχή σε κάθε οργανισμό, σε κάθε φορέα με τον ένα άλλο τρόπο πρέπει να εκπροσωπείται το κοινοβούλιο. Δεν αναφέρθηκα στη μορφή εκπροσώπησης, αυτό το αφήνουμε για αργότερα για διευκρίνηση. Όσον αφορά ενδεχόμενη συγχώνευση αυτών των υπηρεσιών, έχω πολλές θετικές υπηρεσίες, ε, θετικές απόψεις για τις υπηρεσίες. Έχω μεγάλο δυναμικό όσον αφορά την πείρα, όσον αφορά την ε, ε, πρόθεση νέων λύσεων κλπ. το Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να προωθεί τη, φωνή την κοινωνική. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί περνάμε κρίση και δεν υπάρχει μία και μοναδική πανάκια για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής. Άρα, κατά την άποψή μου, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με την κατάρτιση και την κοινωνική πολιτική. Είμαι ανοιχτό για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας να αναλύσουμε το κείμενο μαζί και να συνεργαστούμε τους κοιόδης συγγητέ. Ευχαριστώ. Βασίζομαι σε αυτά τα τελευταία που είπατε. Διότι παρόμοια ανησυχία και εγώ, έχω και εγώ με τη δική σας. Θυμούμε ότι σε κάνα δύο επισκέψεις σε κάποιον από αυτούς τους φορείς διαπίστωσα ότι η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και των φορέων αυτών ήταν ε, πιο περίπλοκη, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει στο πρόγραμμα εργασιών τους. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθα σε επαφή με τον Επίτροπο για να ζητήσω, να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να και λοιπά. Τα ξέρει η κυρία Λαμπέρ που είναι στην διαθεσμική ε, ομάδα που ασχολείται με το έργο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Ίσως επ' αυτού μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω αναλύσεις. Όμως, εκείνοι που διορίζουμε και πρέπει να τοποθετηθούμε επ' αυτόν αύριο, δεν εκπροσωπούν εκεί το Κοινοβούλιο. Ε, είναι παρόντες σαν εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Κοινοβούλιο. Στην αρχή της θητείας του ζητήσαμε εις βάθος. Όταν έπρεπε να ασχοληθώ τη δικασία. Δεν έχουν εντολή την πλευρά μας αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς τους βάζουμε εκεί λόγω της εμπειρίας τους. Αλλά να είναι σημείο επαφής αυτή για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες κλπ. Έστω, ας γίνει έτσι. Αλλά σας λέω για μια ακόμη φορά ότι δεν έχουν εντολή τέτοια δική μας. Ε, δεν μπορούμε να παρεύουμε άμεσα επί του προγράμματος εργασίας. Ε, πρέπει να το συζητήσουμε με τον Επίτροπο. Και έτσι μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε ίσως το πρόγραμμα εργασιών των Επιτροπών. Γι' αυτό ενδιαφέρθηκα για το θέμα, για τον εξή λόγο. Δηλαδή, ότι αποκεντρωμένοι φορείς, λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσία μπορούν να υποστηρίξουν κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Επίκαιρο παράδειγμα. Έκθεση της κυρίας Κορνέλισεν για την τύση έκθεση στην ανάπτυξη. Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε τέτοια έκθεση ε, έχοντας τη συνδρομή των υπηρεσιών αυτών ε, θα πετυχαίναμε προστιθέμενη αξία λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν. Δεν αρκεί να το αναφέρουμε σε μια έκθεση αυτό. Πρέπει να πάμε πιο πέρα, να δούμε αν θα ξαναεξεταστεί ο κανονισμός και αν θα ξεκινήσουμε εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση με τον Επίτροπο. Είμαι σίγουρη όμως ότι σε αυτό το πνεύμα μπορούμε να προχωρήσουμε. Τουλάχιστον αυτό επιθυμώ και εύχομαι. Όσον αφορά την έκθεσή σας, ακολουθούμε ιδιαίτερη διαδικασία λόγω των προθεσμιών των πολύ στενών για αντίδραση. Άρα, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες, αλλά μόνο αγγλιστή. Για πρώτη, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2012 θα εξεταστούν οι τροπολογίες σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας Ιστρασβούργων. την 13η Φεβρουαρίου. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες τις πρωινές. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Αν φάτε και κάτι καλύτερο από ένα σάντουιτς. Και τα ξαναλέμε στις 3. Γεια σας.